Can Ας ξαναρχίσουμε την απογευματινή συνεδρίαση. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι τα τέλη για την ασφάλεια των αερομεταφορών. Έκθεση του κυρίου Λάιτφριντ, ανταλλαγή απόψεων. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η νομοθετική αυτή πρόταση αναφέρεται σε ένα θέμα το οποίο επιφανειακά φαίνεται απλό. Αφορά το γεγονός ότι τα τέλη για την ασφάλεια της ε, αεροπλοείας των ε, αεροπορικών μεταφορών έχουν αυξήθει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Και αυτό είναι ένα τμήμα του κόστους των αεροπορικών συγκοινωνιών που δεν υπόκειται σε ρύθμιση και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη σε επίπεδο ανταγωνισμού για την αεροπορική βιομηχανία, αλλά επίσης μπορεί να οδηγήσει και σε ζημίες προς την κατεύθυνση των καταναλωτών. Η Κομισιόν για αυτούς τους λόγους προβλέπει να ρυθμίσει τα τέλη αυτά τα αερολιμανικά και τα τέλη ασφαλείας με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να είναι διαφανή και να είναι σαφή στους καταναλωτές, αυτό είναι πάρα πολύ βέβαια φιλόδοξο και περιλαμβάνει ορισμένε βασικές αρχές. Καταρχήν πρέπει να βασίζεται στην μη διάκριση. Δεύτερον, να υπάρχουν οι δυνατότητες διαβούλευσης για, το, για τη στάθμιση του τέλους και για τη νομική προσφυγή. Επίσης, σύνδεση του κόστους του αερολιμενικού με το κόστος ασφάλειας. Όλες αυτές είναι αρχές τις οποίες κατά την άποψή μου μπορεί κανείς να υποστηρίξει. Και είναι απόλυτα δια... είναι απόλυτα τεκμηριωμένα αυτά, όπως όμως ήθιστε ο διάβολος υποκρύπτεται μεταξύ των λεπτομεριών. Και συγκεκριμένα στις λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με τη χρηματοδότηση αυτών των μέτρων, γιατί στην Ευρώπη υπάρχει πραγματικά μεγάλη ανάγκη να γίνουν οι απαραίτητε προσαρμογέ στα θέματα τη ασφάλεια. Εγώ λοιπόν με το στόχο αυτό έχω παρουσιάσει ένα εγγράφο εργασία όπου θέτω όλα αυτά τα ζητήματα για την προσοχή των συναδέλφων. Τίθεται φυσικά το ερώτημα αν θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί πράγματι από την Ευρωπαϊκή Ένωση η ασφάλεια, η ασφάλεια με την έννοια της προστασίας των επιβατών, γιατί αυτή είναι μια κλασική αρμοδιότητα των κρατών μελών είναι τμήμα της κυριαρχίας ενός κράτους υποχρέωση να προστατεύει τους πολίτες του από πιθανούς κινδύνους. Η άλλη πλευρά βέβαια είναι ότι ο αεροπορικός κλάδος είναι ένας τομέας όπου ισχύει πάντα η αρχή ότι ο χρήστης καταβάλει το τέλος. Ο, ο καταναλωτής, ο χρήστης είναι αυτός ο οποίος πληρώνει, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ένα καταλογισμό του κόστου στον καταναλωτή. Όπω βλέπετε αυτή είναι μια τελείω διαφορετική προσέγγιση από την προσέγγιση ότι η ασφάλεια είναι μονάχα υπόθεση του κράτου. Και εδώ θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να διαιτητεύσουμε μεταξύ των δύο αυτό, αυτών απόψεων. Ένα δεύτερο ερώτημα είναι πώς θα καθορίσουμε το ύψος των τελών ασφαλείας. Τι είναι δικαιολογημένο και τι δεν είναι δικαιολογημένο. Και πού εμπλέκεται η αρχή ότι ο χρήστη θα πρέπει να πληρώνει. Και υπάρχει μια πρόταση από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που κινείται προς την κατεύθυνση που λέει ότι θα πρέπει να υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνες οι οποίοι θα δίνουν γενικές λύσεις αν κάποια κρατημέλη θέλουν να εξασφαλίσουν ένα υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί χρηματοδοτικά από τα ίδια τα κρατημέλη. Και μπορεί κανείς να προβλέψει λοιπόν τη δυνατότητα να υπάρχει μια διαφοροποιημένη παροχή ασφαλής υπάρχει μια τρίτη παραλλαγή η οποία δεν ασχολείται καθόλου με το θέμα του ποιος θα πληρώνει τελικά το κόστος, απλώς θέλει να υπάρξει μια ισοδίκια κατανομή του κόστους. Το τελευταίο ερώτημα είναι το κατά πόσον η ασφάλεια των πτήσεων, η ασφάλεια των αεροπορικών συνδέσεων θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο εφόσον ρυθμίζεται πια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι το οποίο θα σήμαινε θα πρέπει να δοθούν ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα για την εξασφάλιση της ασφάλειας. Αυτές είναι οι βασικές επιλογές λοιπόν για την χρηματοδότηση. Εμείς πιστεύω θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση επί της ουσίας για τα θέματα αυτά. Βέβαια, εγώ δεν έχω κάποια συγκεκριμένη προτίμηση μεταξύ των επιλογών που διέγραψα προηγουμένως. Θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η άποψη των συναδέλφων από τις διάφορες πολιτικές ομάδες και θα ήθελα ή δυνατόν στις παρεμβάσεις των συναδέλφων να ακούσω τις απόψεις τους για το πώς θα έπρεπε να ρυθμιστεί το θέμα της χρηματοδότησης. Είναι χρήσιμο λοιπόν να σκεφτούμε για το θέμα αυτό γιατί βρισκόμαστε ενώπιον μιας κατάστασης όπου υπάρχει δυνατότητα να παραταθεί η, η ρύθμιση για τα υγρά, για τη μεταφορά των υγρών, να χρησιμοποιηθούν νέες συσκευές οι οποίες κοστίζουν 200 ευρώ τουλάχιστον το κομμάτι. Για να εγκατασταθούν λοιπόν αυτές οι συσκευές κάποιος πρέπει να πληρώσει. Το ερώτημα είναι πώς θα κατανεμηθεί το κόστος αυτή, αυτών των εγκαταστάσεων. Και αυτό είναι ένα από τα ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και επίσης πιστεύω ότι αυτή η οδηγία δεν έχει λάβει υπόψη επαρκώς το θέμα της προστασίας του καταναλωτή δεν έχει αυτή την προβληματική αντιμετωπίσει επαρκώ και θα πρέπει να κάνουμε κάτι σε σχέση με αυτό. Υπάρχει επίσης το θέμα του πώς καθορίζουμε, πώς ορίζουμε την ε, έννοια του τέλους ασφαλείας. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά βελτιώσιμη η πρόταση της Κομισιόν, η διατύπωσή της για το θέμα αυτό. Όλα αυτά όμως βέβαια δεν είναι τα θέματα ουσίας. Το θέμα της ουσίας είναι πώς θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν όλα αυτά τα μέτρα και επίσης θα πρέπει να καταλήξουμε και σε μερικές βασικές αρχές, και εδώ θα κλείσω. Θα πρέπει να βρούμε ένα υπόδειγμα, ένα τρόπο ρύθμισης που να λαμβάνει υπόψη ορισμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, το ότι υπάρχουν ήδη υποδείγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα οποία λειτουργούν ικανοποιητικά, λειτουργούν γενικά προς την κατεύθυνση της ικανοποίησης των περισσότερων χρηστών και δεν πρέπει να έχουμε μία ρύθμιση η οποία θα εμποδίσει τέτοιου είδου υποδείγματα να λειτουργούν και στο μέλλον. Αντίθετα, θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να συνεχίσει τη λειτουργία τους. Δεύτερον, δεν θα πρέπει και δεν θέλουμε εξάλλου να αφαιρέσουμε την ευθύνη των κρατών μελών και την αρμόδιότητά τους για το τι είναι απαραίτητο μέτρο ασφάλειας και το τι δεν είναι. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να μείνει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, τι επίπεδο ασφάλειας θέλουν να εξασφαλίσουν στους πολίτες και τι επομένως δαπάνες είναι έτοιμα να δώσουν προς την κατεύθυνση της ασφάλειας. Αυτό όμως το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιο μοντέλο χρηματοδότησης. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε τελείως στην διακριτική ευχαίρεια των κατώμελων. Δηλαδή Τρίτον, υπάρχουν ορισμένες εξελίξεις οι οποίες δεν είναι πάντα θετικές. Θα πρέπει να αποφύγουμε σφάλματα και δημιουργία κενών, θα πρέπει να έχουμε μία αντιμετώπιση η οποία θα εξασφαλίσει ότι όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να γίνουν δεν θα είναι κατά ανάγκη πολυδάπανα. Δηλαδή να βρούμε έναν τρόπο να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει εξέλιξη στον τομέα αυτό και να μην εμποδίσουμε την εξέλιξη της τεχνολογίας για τον τομέα αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν σε μια συζήτηση η οποία για μένα τουλάχιστον είναι συναρπαστική. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Lightfoot. εκπρόσωποι των ομάδων. Ασάδα από το ΕΛΚ. ο πρώτος αγορητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε, λέει και ο Ζασάντα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε. Διάβασα προσεκτικά το έγγραφό του, το οποίο εμπεριέχει αρκετά ενδιαφέρουσες προτάσεις, οι οποίες με έπεισαν να ετοιμάσω διάφορες ε, προτάσεις σχετικά με το τι μπορεί να γίνει παραπάνω με το έγγραφο. Το θέμα της ασφαλείας, κυρίως μετά την 11η ε, Σεπτεμβρίου, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για μένα προσωπικά, όπως και για άλλους ταξιδιώτες που χρησιμοποιούν τις αεροπορικές εταιρείες είναι πολύ πιο κρίσιμο θέμα από την άνεση των πτήσεων. Ε, Ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που είπε ο εισηγητής και να υπογραμμίσω κάποια πράγματα. Το πιο σημαντικό ζήτημα είναι η χρηματοδότηση και η Επιτροπή βέβαια κατέληξε σε τέσσερις προτάσεις και μία από αυτές ε, θέλει να καταλήξουμε σε ένα πλαίσιο εντός του οποίου θα καθορίσουμε τα τέλη. Αυτό που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το κράτος να φέρει την ευθύνη για την ασφάλεια και να χρηματοδοτεί την ασφάλεια. Εγώ υπογράμμισα κάποια σημεία του κειμένου στην έκθεση όπου αναφέρεται, όπου φαίνεται ότι αποφεύγει να αντιμετωπίσει κατευθείαν το θέμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρόλο που ε, τελικά αξιολογεί θετικά τη χρηματοδότηση ασφάλειας από πλευράς κράτους. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να πληρώνουν εκείνοι που δεν ταξιδεύουν. Να μην πληρώνουν δύο φορές. Πληρώνουν καταρχάς φόρους. Δεν πρέπει να πληρώνουν και δεύτερη φορά, εφόσον δεν χρησιμοποιούν τα αεροπλάνα δεν θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι που δεν πετάνε να πληρώνουν για την ασφάλεια. Εκείνοι που είναι επιβάτες πληρώνουν δύο φορές. Πληρώνουν και αυτοί φόρους και μετά πληρώνουν και το κόστος της ασφάλειας, διότι δεν χρηματοδοτείται συνολικά το κόστος από το κράτος. Ούτε από τις αεροπορικές εταιρείε, αλλά από τους επιβάτες. Εκείνοι είναι που τελικά πληρώνουν το τίμημα. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ εκείνων των επιβατών και εκείνων των ανθρώπων που ταξιδεύουν με τρένο, που ταξιδεύουν με το αυτοκίνητο. Εν τη αυτή περιπτώση φροντίζει για την ασφάλειά τους το κράτος. Το κράτος χρηματοδοτεί την ασφάλεια όσον αφορά τις δημόσιες μεταφορές και υπάρχουν φορείς που ελέγχουν αν υπάρχει αυτή η ασφάλεια. Εκείνοι λοιπόν που χρησιμοποιούν άλλες ε, μορφές μεταφορών δεν χρειάζεται να πληρώνουν παραπάνω χρήματα ή την ασφάλεια. Το κράτος τους προστατεύει προστατεύει και τους ανθρώπους στα σημεία ε, διελεύσεως των συνόρων. Δεν επιτρέπει σε επικίνδυνα άτομα να μπουν στη χώρα με διάφορες ουσίες, που ίσως ουσίες αυτές να είναι επικίνδυνες. Δεν βλέπω λοιπόν γιατί οι επιβάτες των αεροπλάνων να αποτελούν αντικείμενο διάκρισης πληρώντας δύο φορές. Πληρώνουν και φόρο και πληρώνουν και μία επιβάρυνση πάνω από την τιμή του Εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή ότι το Συμβούλιο ίσως να απορρίψει μια τέτοια λύση. Και θα ήθελα να υποστηρίξω ένα μεικτό σύστημα. Ένα τμήμα του κόστους καταβάλλεται από το κράτος και ένα άλλο τμήμα του κόστους καταβάλλεται από τα αεροδρόμια και τις αεροπορικές εταιρείες. Πρέπει να έχουμε όμως υπόψη ότι τελικά θα την πληρώσουν οι επιβάτες. Στην τρίτη πρόταση, ο κύριος εισηγητής πρότεινε να μην εξεταστεί το θέμα της χρηματοδοτήσεως, παρόλο που πιστεύω ότι θα επανέλθει σαν μπούμεραγκ αυτό το θέμα. Αν δεν το πιάσουμε σήμερα, θα το πιάσουμε κάποια άλλη φορά στο μέλλον. και είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Αναρωτιέμαι πώς ποσοστιαία θα υπολογίσουμε το μερίδιο, το μερτικό του κράτους. Η διαδικασία του υπολογισμού του κόστους, του λεπτομερούς υπολογισμού του κόστους, ε, είναι κάτι αρκετά περίπλοκο. Πρέπει να υπολογίσουμε πρώτα το κόστος. Και είναι περιπλοκότατη αυτή η διαδικασία. Και κοστίζει και αυτή η διαδικασία υπολογισμού του κόστους. και γι' αυτό θα πρέπει να αυξηθούν ακόμα περισσότερο τα τέλη. Και έχω άλλες δύο προτάσεις, άλλα δύο θέματα που θέλω να θίξω. Αν τα τέλη επιβληθούν από τις αεροπορικές εταιρείες υπό την εποπτεία κάποιας αρμόδιας αρχής που θα δημιουργηθεί, κάτι που βέβαια πάλι προσθέτει στο συνολικό τόξο, ε, κόστος, συγγνώμη, τότε διαρωτώ με, τι θα κάνουν τα αεροδρόμια. Θα μειώσουν το κόστος λόγω ανταγωνισμού. Λόγω ανταγωνισμού μεταξύ αεροδρομίων, μήπως τελικά υποτιμήσουν το κόστος εις βάρος της ασφάλειας των επιβατών. Από την άλλη, ίσως να αυξήσουν τα τέλη, τα αεροδρόμια, εκεί όπου δεν φοβούνται τα αεροδρόμια τον ανταγωνισμό μεταξύ αεροδρομίων. για να αντισταθμίσουν τις συνέπειες της κρίσης και για να συμπληρώσουν τον προϋπολογισμό τους. Και ένα ερώτημα έχω τώρα που απευθύνω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς προτίθεται να καταστήσει το κόστος διαφανές. Ελπίζω να μπορείτε να μου απαντήσετε. Και σαν εκπρόσωπος της ομάδας μου, ελπίζω να μπορέσω να παρακολουθήσω από κοντά τη συζήτηση και εκτιμώ τη δυνατότητα που είχα να εκφράσω τις απόψεις μου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σαν τεζαβού είναι αυτό για μας, όσοι είμαστε εδώ και ήμασταν στο, στην παλιά θητεία. Ήταν ενδιαφέρον να ξανακούμε αυτά που υπόθηκαν. S&D, κύριος Αλκαντράουι έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον ε, εισηγητή. Πραγματικά, πολύ καλά τα λέει και ειδικότερα ως προς τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι κάτι καινούριο. Από τον ε, πρώτο κανονισμό του 2001, εμείς ως Κοινοβούλιο πάντοτε θέλαμε να είναι απολύτως σαφές πώς ε, πληρώνονται τα τέλη ασφαλείας. Μα είχε υποσχεθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα μα υποβάλει πρόταση, αλλά δεν είδαμε τίποτε τέτοιο. Η αναθεώρηση της οδηγίας ε, οδήγησε σε μια νέα οδηγία το 2008 και ούτε εκεί καταφέραμε να πάρουμε αυτό που θέλαμε. Και τώρα μιλούμε ήδη για μια καινούργια πρόταση. Δύο σημαντικά ζητήματα θα ήθελα να θέσω και που πρέπει να τα λύσουμε. Πρώτον είναι το θέμα της διαφάνειας. η διαφάνεια για τον κλάδο, για τους εμπλεκομένους φορείς, ε, αλλά και για τους χρήστες, για τους καταναλωτές. Και τι εννοώ με αυτό. Ότι πρέπει να μπορεί ο καθένας να γνωρίζει τι ακριβώς πληρώνει και, αυτό, και ότι αυτό για το οποίο πληρώνει χρησιμοποιείται πράγματι για τη βελτίωση της ασφάλειας. Αυτό είναι πολύ σημαντική πτυχή της ασφάλειας. Για παράδειγμα, αν, θα υπάρξει όντως, ε, αν υπάρξει όντως τέλος ασφαλείας, ε, τα χρήματα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ε, για νέες θέσεις, πάρκινγκ για παράδειγμα. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και, συνεφο, και συνεπώς πρέπει να υπάρξει και σωστή διαβούλευση. Το δεύτερο θέμα είναι ποιος θα πληρώσει την ύφη. Ποιος θα αναλάβει το κόστος. Το Κοινοβούλιο πάντοτε θεωρούσε ότι πρέπει να υπάρξει μια διάκριση μεταξύ των μέτρων ασφαλείας που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο ε, Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που είναι αρμόδια για την υποβολή προτάσεων για το θέμα αυτό και από την άλλη υπάρχουν και τα επιπρόσθετα μέτρα τα οποία θέλει, θέλουν τα κράτη-μέλη να ε, λάβουν επιπλέον. Αυτό που νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουμε είναι μεικτή χρηματοδότηση. Μεικτή χρηματοδότηση ώστε και ο κλάδος και οι καταναλωτές να συμμετέχουν ε, στη, στα τέλη αυτά. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να αποφασίσουμε πρέπει να είναι σαφές σε κάθε, ε, σε κάθε ένα ποιος πληρώνει τι. Τώρα τα επιπλέον μέτρα που θέλουν ε, να λάβουν τα κράτη-μέλη εκτός από τα ευρωπαϊκά μέτρα, κοιτάξτε, εγώ ξεκινώ από την υπόθεση ότι τα ευρωπαϊκά μέτρα κανονικά θα πρέπει να αρκούν για την ασφάλεια, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν τα κράτη-μέλη θέλουν επιπρόσθετα μέτρα, πρέπει να δεχθούν και μία, να αναλάβουν μια να λάβουν οικονομική ευθύνη. Αυτό που νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε είναι να αναπτύξουμε ένα σύστημα που εξασφαλίζει ότι οι υπεύθυνοι για την ασφάλεια ενθαρρύνονται να σκεφτούν τις συνέπειες όλων όσων κάνουν. Δεν θα έπρεπε απλώς να συσσωρεύονται τα μέτρα ασφαλείας το ένα πάνω από το άλλο Είδαμε πώς, έχουν αυξηθεί, πώς έχει αυξηθεί το κόστος ε, γενικώ. ...35% περίπου είναι τα τέλη, το επιπλέον κόστος λόγω των ε, επιπλέον μέτρων ασφαλείας... ...και είναι πολύ μεγάλο το κόστος αυτό για να μην είναι σαφή τα πράγματα και για να μην υπάρχει διαφάνεια. Πρέπει να ξέρουμε ακριβώς για τι μέτρα μιλάμε και ποιος πληρώνει για αυτά τα μέτρα. Και μία ακόμη ερώτηση, η κοινοτική χρηματοδότηση χρειάζεται? Σε σχέση με τη συζήτηση για τα υγρά ε, εντός των ε, αεροσκαφών, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι θα αναλάβει τη χρηματοδότηση διαφόρων δοκιμών. Εγώ νομίζω ότι αν δεν υπάρχει επιπλέον κοινοτική χρηματοδότηση, Δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτήσουμε όλα αυτά τα νέα συστήματα ασφαλείας, αλλά υποθέτω ότι αν δεν θέλουμε να υπάρξουν αλλαγέ στι δημοσιονομικέ προοπτικέ, δεν, δεν είναι δυνατόν να μην κάνουμε επιλογέ. Πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε και μια επιλογή. Κυρία Χάνη Πλασάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ έχω το ίδιο πρόβλημα με εσάς νιώθω μια κόποση γιατί είναι κάτι το, ένα έργο που το έχουμε ξαναδεί. Ξεκινώντας με τον κανονισμό 23-20 με κουράζει το γεγονός ότι και πάλι είμαστε υποχρεωμένοι να επιληθούμε για το ίδιο θέμα. Αλλά ο στόχος μας θα πρέπει να είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι χρήστες θα είναι πλήρως πληροφορημένοι για τον τρόπο με τον οποίο οργανώνται τα μέτρα ασφάλειας που φυσικά θα πρέπει να γίνει αυτό με έναν τρόπο ο οποίος είναι διάφανος τα μέτρα ασφαλείας θα πρέπει να βρίσκονται να υπάρχει σύνδεση του κόστους με τα μέτρα ασφαλείας, θα πρέπει να είναι συνεκτικά τα μέτρα αυτά και να έχουν σαν πραγματικό στόχο να αυξήσουν την ασφάλεια. Και αυτό ισχύει και με τα υγρά τα οποία μεταφέρονται φυσικά. Κάτι ακόμα. Η... Το έγγραφο του εισηγητή λέει ότι θα πρέπει να σκεφτούμε και ποιος θα πληρώσει τι. Αυτό με με οδηγεί να σκεφτώ το εξή. Η Κομισιόν δεν λέει απολύτω τίποτα σε σχέση με τι κρατικέ επιδοτήσει, κάτι το οποίο είναι υποσυζήτηση εδώ και πολύ καιρό. Και η ομάδα μου, η ομάδα των φιλελευθέρων, ήδη έχουν, ε, έχει προσελκύσει αυτό το θέμα την προσοχή μας, ίσως και οι άλλες πολιτικές ομάδες σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο. Μπορούν να υπάρχουν βέβαια διαφορέ μεταξύ των κρατών μελών, αλλά θα πρέπει να γίνει αυτό μέσα στα πλαίσια τη διαφάνεια, πιστεύουμε. Φανταστείτε όμω ένα κράτο το οποίο επομίζεται ένα μεγάλο μέρο του κόστου ασφάλεια για πτήσει οι οποίε πηγαίνουν σε ένα άλλο κράτο μέλο, το οποίο από τη δική του πλευρά δεν δίνει μια τέτοια επιδότηση για την ασφάλεια. Αυτό οδηγεί σε μια κάποια έλλειψη ισορροπία και έλλειψη δικαιοσύνη. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει μέσα στην Ευρώπη. Γι' αυτό δεν μπορούμε να έχουμε μια τέτοια επιλεκτική αντιμετώπιση. Γι' αυτό τονίζω ότι για την ομάδα των φιλελευθέρων είναι απαραίτητο να είναι σαφεί οι αρχέ για το ποιο πληρώνει πότε και πού και κάτω από ποιε προποθέσει επομένω. Και εγώ δεν συμφωνώ να υπάρξει μια κοινοτική χρηματοδότηση ή μια συγχρηματοδότηση, γιατί πάντα ένα τμήμα αυτή τη χρηματοδότηση θα έρθει από τα κάτι μέλη, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ισότητα μεταχείριση των αεροδρομίων. Ευχαριστώ κυρία Φώστερ από το Κόμμα των Συντηρητικών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τον κύριο Λάιχτφριντ για τον τρόπο με τον οποίο έχει διεξαγάγει συζητήσει με του χειώδει συζητητέ σε σχέση με την έκθεση αυτή. Επειδή ήμουν στο παρελθόν εισηγήτρια για το 2320 και εγώ βρίσκομαι στα πλαίσια του Deja Vu, και θυμάμαι και πάλι τι συζητήσει που είχαν γίνει τότε για τη χρηματοδότηση. Αν επιστρέψουμε στην αρχική συζήτηση που ξεκίνησε ουσιαστικά μετά την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, τα βασικά θέματα τα οποία θέσαμε δεν ήταν το αν θα πρέπει τα κράτη-μέλη να πληρώσουν το σύνολο τη χρηματοδότηση ασφάλεια και το θυμόσαστε εσεί κύριε Πρόεδρε, γιατί και εσεί είσαστε παρόν και ιδιαίτερα ενεργό για το θέμα αυτό. Αυτό το οποίο ελέγχθη τότε και υποστηρίχθηκε από την Κομισιόν και υποστηρίχθηκε από την Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ότι το πρόσθετο κόστος ασφάλειας μετά την 11η Σεπτεμβρίου, το οποίο επομίζονται οι αεροπορικές εταιρείες και ο καταναλωτής, ήταν τεράστιο. Σε τελική ανάλυση, ο καταναλωτής πληρώνει, γιατί όλο το κόστος μετακυλίζεται τελικά στον καταναλωτή. Και οι αεροπορικές εταιρείες το κάνουν αυτό, πληρώνουν και αυτές. Αλλά θεωρήσαμε ότι επειδή η απειλή της τρομοκρατίας στρέφεται όχι εναντίον ενός πολίτη ή εναντίον μιας αεροπορικής εταιρείας που είναι απλώς ένα εργαλείο, στρέφεται εναντίον ενός κράτους και η απειλή της τρομοκρατίας στρέφεται εναντίον των κρατών, θεωρούμε ότι το κάθε κράτος έχει μία <clears throat> υποχρέωση να αρρωγήσει τις εταιρείε να αντιμετωπίσουν αυτό το αυξανόμενο κόστος. Όχι να πληρώσει το κόστος, αλλά να βοηθήσει τις εταιρείε να απομισθούν αυτό το πρόσθετο κόστος για τις εταιρείε και τον καταναλωτή. Συμφωνήσαμε τότε ότι αυτό πρέπει να κάνουμε. Ξέραμε ότι ήταν πολύ δύσκολο, γιατί <clears throat> δεν ζητούσαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάτι τέτοιο και η απόφαση να μην υποστηρίξουμε χρηματοδοτικά τα αυτές τις ενέργειες δεν, ήταν απόφαση της Κομισιόν. <clears throat> Και δεν ήταν τα μέλη της δικής μας Επιτροπής που διαφώνησαν. Το Συμβούλιο ήταν αυτό που εμπόδισε αυτές τις <clears throat> προσπάθειες γιατί φάνηκε ότι τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να βάλουν καθόλου το χέρι στη τσέπη για οποιοδήποτε από τμήμα αυτού του πρόσθετου κόστους που έχουμε επομιστεί όλοι ως καταναλωτές. Ελπίζω λοιπόν ότι θα γίνει κατανοητή η θέση μας και η θέση του Μπραντ Σίμψον, ο οποίος είναι πρόεδρος σήμερα. Δεν λοιπόν πρέπει να σταματήσουμε να τονίσουμε ότι υπάρχει έλλειψη δικαιοσύνης σε αυτή την περίπτωση και θα πρέπει να υπάρξει και κάποια υποστήριξη από τα κράτη-μέλη, γιατί στο σημερινό καθεστώς ο καταναλωτής τα πληρώνει όλα. Αυτά λοιπόν για την υπόθεση της χρηματοδότησης. Είναι λιγάκι διαφορετικά από αυτά που λέει ο κ. Λάιχτφριντ στο εγγραφό του, που έχει μια κάπως διαφορετική προσέγγιση. Αλλά η προσέγγιση του κ. Λάιχτφριντ αφορά την οδηγία για τα αερολιμενικά τέλη. Εγώ δεν ενεπλάκην σε αυτό το θέμα, παρά το γεγονός ότι το παρακολούθησα από μια άλλη οπτική γωνία. Προφανώς λοιπόν όλα αυτά τα θέματα μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Αλλά το θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να κατανοήσουμε περί τίνος πρόκειται. Δεν μπορούν όλα αυτά τα θέματα να θεωρηθούν ότι είναι αερολιμανικά τέλη, γιατί το κόστος της ασφάλειας είναι ένα πολύ πιο πολύπλοκο πρόβλημα. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε ένα τρόπο πιο ήπιο να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Αυτά τα οποία κάναμε εμείς μετά την 11η Σεπτεμβρίου ήταν να ζητήσουμε από τα τότε 15 κράτη-μέλη να μας πούν με ποιο τρόπο κατανέμαν και καταλόγησαν το κόστος ασφάλειας. Κάποια κράτη-μέλη πληρώναν ένα τμήμα αυτού του πρόσθετου κόστους, αλλά όχι. Τώρα όμως έχουμε 27 κρατη 27 διαφορετικές μεθόδους χρηματοδότησης. Μερικά μπορεί να καλύπτουν το κόστος των αστυνομικών που περιπολούν στα αεροδρόμια. Άλλοι, όπω το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν το κάνουν. Λένε ότι αυτό πρέπει να το πληρώσει ο καταναλωτή. Δεν νομίζω ότι μπορούμε εμεί να τα καταλύσουμε αυτά και να γυρίσουμε στο status quo άντε πριν από την 11η Σεπτεμβρίου. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Απλώ θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το ότι όλα αυτά είναι ανοιχτά και διάφανα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν τεράστιες διαφωνίες εδώ μεταξύ αυτών που εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση, αλλά ξέρουμε ότι τα αεροδρόμια και οι καταναλωτές θα πρέπει να συζητούν πιο συχνά για τα θέματα αυτά και να υπάρξει κάποιος τρόπος να καθορίσουν αυτά τα τέλη. Αυτή είναι μια πιο σιωπηλή μέθοδος, η οποία όμως λειτουργεί. <clears throat> αλλά εγώ δεν έχω πάρει μια θέση σε αυτή τη διαφωνία μεταξύ των καταναλωτών και των αεροδρομίων. Είναι τεράστιες οι διαφορές απόψε μεταξύ τους. Τα αεροδρόμια λένε δεν σας χρεώνουμε αρκετά, οι καταναλωτέ λένε μα χρεώνεται πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό το οποίο δεν πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να παίξουμε το ρόλο του διαιτητή μεταξύ των δύο αυτών πλευρών. Όσο και να του αγαπώ και του μεν και του δε. Δεν είναι αυτό ο ρόλο μα. Αυτό το οποίο προτείνω είναι να έχουμε εθνικέ ρυθμιστικέ αρχέ, τι αρχέ πολιτικέ αεροπορίε, οι οποίε υπάρχουν ήδη και θα πρέπει να εξετάσουμε με ποιο τρόπο τα αεροδρόμια και οι αεροπορικές εταιρείες χρησιμοποιούν τις εθνικές βοήθειες. Αν υπάρξει μια διαφωνία μεταξύ των αεροπορικών εταιρείων και των εταιρείων και των αεροδρομίων, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν οι συζητήσει για τα θέματα αυτά και να υποχρεώσουμε τι δύο πλευρέ να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Δεν χρειαζόμαστε ένα κανονισμό να το κάνουμε αυτό. Γιατί ήδη θα έπρεπε οι δύο πλευρέ να έχουν συμφωνήσει για το πώ θα κάνουμε όλα αυτά και δεν πρέπει εμεί να παίξουμε ένα διαιτητικό ρόλο. Εν κατακλείδη λοιπόν. Νομίζω ότι ο κ. Λάχτφριντ έχει ακολουθήσει μια σωστή προσέγγιση. Δεν θέλουμε εμεί σαν Επιτροπή να περιπλέξουμε ακόμα περισσότερο αυτό το θέμα. Δεν θέλουμε να καταλύσουμε τι συμφωνίε οι οποίε έχουν επέλθει. Δεν θέλουμε, ανεξάρτητα από το τι θα προκύψει, να κάνουμε κάτι το οποίο θα δώσει ακόμα μεγαλύτερο βάρος στον καταναλωτή, θα αυξήσει το κόστος των ναύλων από τον καταναλωτή. Νομίζω ότι ήδη είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια και είναι υψηλό το πρόσθετο τέλος που πληρώνουμε για την ασφάλεια, εγώ υποθέτω ότι όλα αυτά τα χρήματα χρησιμοποιούνται για το σωστό σκοπό μέχρι αποδείξεις του αντιθέτου. Αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε μια σαφή θέση ως Επιτροπή Μεταφορών. Ο κύριος Δεγράνδες Πασκουάλ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βρισκόμαστε σε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Και βλέπω να επαναλαμβάνεται η διαφορά απόψεων και οι λόγοι, η αντιμετώπιση, τα επιχειρήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν. Το βασικό πρόβλημα <clears throat> δεν είναι η αξία της προστασίας και η αξία της ασφαλείας στα αεροδρόμια και στις πτήσεις. Το βασικό θέμα είναι η ουσία, δεν είναι οι λεπτομέρειες. Η ουσία είναι το ποιος τις πληρώνει, ποιος θα φέρει το κόστος της ασφάλειας. Εγώ πιστεύω ότι ήταν ισορροπημένη και η θέση του εισηγητή και των σκιωδών εισηγητών. Από τη στιγμή που θα κατατεθεί το έγγραφο εργασίας η, μάλλον η έκθεση του εισηγητή, μπορούμε να καταθέσουμε τροπολογίες και να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε κάποια κοινή θέση. Η ασφάλεια δεν είναι ένα μικρό θέμα, μια λεπτομέρεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα η ασφάλεια. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή υπάρχει και μια τεράστια υποστήριξη από τους πολίτες για να εξασφαλιστεί παστησία ή ασφάλεια. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε αν αυτή η ασφάλεια πρέπει να εξασφαλίσεται από τις αεροπορικές εταιρείε ή από το κράτος. Να δούμε λοιπόν ποιος είναι αυτός ο οποίος πληρώνει την ύφη αυτής της μεγάλης αξίας που είναι η ασφάλεια. Αυτή είναι μια πολύ παλιά συζήτηση. Η ισπανική θέση στο Συμβούλιο, και το λέω αυτό <clears throat> γιατί η αντιμετώπιση αυτής της οδηγίας θα συμπέσει ουσιαστικά με την Ισπανική Προεδρία, η άποψη της Ισπανίας είναι ότι αυτό το κόστος πρέπει να το επομίζεται ο προϋπολογισμός της κάθε χώρας. Ότι δεν πρέπει, συγγνώμη, να το κάλυπτει ο γενικός προϋπολογισμός, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα τέλη τα οποία θα πληρώνει ο χρήστης. Αυτό ίσως είναι πολύ δραστικό για ορισμένους οι οποίοι δεν έχουν δοκιμάσει ένα τέτοιο σύστημα. Αλλά πιστεύω ότι η καλύτερη λύση είναι να υπάρχει ένα μεικτό σύστημα το οποίο θα εξασφαλίσει μια ισορροπία. Προφανώς ο καταναλωτής θα πρέπει να υπομειστεί ένα τμήμα αυτού του κόστους, αλλά όχι το σύνολο. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια συζήτηση μεταξύ μας για να δούμε πώς θα μπορέσει να υπάρξει μια καταρμή του κόστους μεταξύ κράτους και καταναλωτών. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Ντιγκράνης Πασκάλ. Ο κύριος Λιμπεράτσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι συμφωνώ αρκετά με την κυρία Φώστερ η οποία είπε ότι εμείς δεν, δεν θέλουμε να προστατεύσουμε τις εταιρείε θέλουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες όταν οι τρομοκράτες θέλουν να χρησιμοποιούν τι αερομεταφορέ κατά αυτόν. Λοιπόν, αυτό πάντα το έχουμε υπόψη. Όταν είδαμε τι έγινε στο, στα γεγονότα της Νέας Υόρκης 11 Σεπτεμβρίου και το πώς χρησιμοποιήθηκαν, τι αξία είχαν τα αεροπλάνα που χρησιμοποιήθηκαν στα εργαλεία, δεν ήταν πολύ ακριβά εργαλεία. Δεν μιλάμε για τον τομέα των αερομεταφορών και την ασφάλεια των αερομεταφορών, μιλάμε για την ασφάλεια των πολιτών, την ασφάλεια των ανθρώπων. Έχουμε διάφορους αερολιμένες, διαφορετικούς. Ας πάρουμε το, το Heathrow ή το Stetsin στην Πολωνία. Η δυνατότητα να έχουν εξοπλισμό ασφαλείας. Για να κάνουν τη δουλειά τους και υποτίμηση η απαξίωση του εξοπλισμού έχουν διαφορετικά ποσοστά για το Στέτσιν και για το Heathrow. Αλλά υποτίθεται ότι τα αποτελέσματα πρέπει να είναι τα ίδια. Επίση, διαφέρει η κατάσταση στο ποιο φροντίζει για την ασφάλεια. Έχουμε αστυνομικού, έχουμε τολωνιακούς, έχουμε ιδιωτικέ ε, εταιρείε ασφαλεία που προσλαμβάνονται από τα αεροδρόμια. Οπότε ποικίλει η κατάσταση από αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο. Μεγάλε διαφορέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο εισηγητής ε, έκανε πολύ καλή δουλειά, έδωσε επιλογές και έδωσε δυνατότητες δράσης και μας καλεί όλους να συζητήσουμε. Θα ήθελα ακριβώς γι' αυτό να τον ευχαριστήσω. Από ό,τι καταλαβαίνω θέλουμε να έχουμε ε, εναρμονισμένους κανόνες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ανταγωνισμός και η λειτουργία και ο επιμερισμός του βάρους στον τομέα αυτό θα πρέπει να είναι συγκρίσιμα στοιχεία σε όλα τα κράτη-μέλη. Τέλος πάντων, δεν πρέπει να τσακωνόμαστε εμείς και οι πολίτες θα πληρώσουν. Το θέμα είναι αν η πληρωμή θα γίνει έμεσα μέσω φορολόγησης, φόρου που πάει στο κράτος, ή άμεσα αν θα πληρώσουμε το τίμημα ως επιβάτες που θέλουμε να επιβιβαστούμε σε ένα αεροσκάφος. Αν θέλουμε να έχουμε συγκρίσιμες συνθήκες και λάβουμε υπόψη τι γίνεται σε άλλους τομείς, θα πρέπει να επιλέξουμε ένα μεικτό σύστημα. Στο μεικτό σύστημα ο κρατικός τομέας και ο ιδιωτικός τομέας συμπεριλαμβάνονται. Γιατί χρειαζόμαστε το κρατικό σύστημα, το δημόσιο σύστημα. Το χρειαζόμαστε διότι μιλάμε για ασφάλεια με την ευρύτερη έννοια του όρου. Δεν μιλάμε μόνο για την προστασία και την ασφάλεια των επιβατών μέσα στο αεροσκάφο, αλλά μιλάμε για πολλά περισσότερα όσον αφορά την ασφάλεια. Χρειαζόμαστε αεροδρόμια, αεροπορικέ εταιρείε και το κρατικό σύστημα να συνεργαστούν όλοι οι τομείς για την ασφάλεια, γιατί έτσι είναι πιο εύκολο να πετύχουμε το σωστό διάλογο και να καθορίσουμε διατάξεις και προδιαγραφές όσον αφορά την οικονομική ευθύνη. Νομίζω ότι οι ρυθμιστικές αρχές δεν θα πρέπει να ρυθμίζουν την κατάσταση μόνο για εκείνους που πληρώνουν για τη θέσπιση των ρυθμίσεων. Συμφωνώ με εκείνους που λέγουν ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είναι αόρατη εν τη αυτή περιπτώση και δεν γνωρίζουμε γιατί θα έπρεπε και αυτός ο φορέας να συμμετάσχει και να επομιστεί τις ευθύνες του. Ενθαρρύνω λοιπόν αυτό το φορέα, αυτή την υπηρεσία να κάνει ακριβώς αυτό και ενθαρρύνω και μας να πλησιάσουμε ολιστικά το θέμα. Να μην διατηνόμεθα ότι προστατεύουμε μόνο τις αεροπορικές εταιρείες, προστατεύουμε όλους μας, όχι μόνο τις αερομεταφορές και μακροπρόθεσμα θέλουμε να αποθαρρύνουμε εκείνους που θέλουν να ασκήσουν τρομοκρατία και θέλουν να απειλήσουν την ασφάλεια ε, από πολλές πτυχές, δηλαδή να απειλήσουν την ασφάλεια εκ πλευράς οικονομικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ο κ. Bradburn. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βέβαια, είχε δίκιο η κυρία Φώστερ σε αυτά που είπε και μας υπενθύμησε και τη συζήτηση που είχαμε κάνει στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία όταν ε, ασχοληθήκαμε με την πρόταση της ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας. Δηλαδή, θα θυμάστε κι εσείς, ε, κάποιοι συνάδελφοι ήταν και τότε παρόντες, ότι υπήρξαν διαπραγματεύσεις ε, στο προηγούμενο κοινοβούλιο για να μπορέσουμε να επιτύχουμε μια συμφωνία επί της πρότασεως. Φτάσαμε στην συνδιαλλαγή και θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους σας ότι ένα ζήτημα που δεν επιλύσαμε κατά τη διάρκεια της συνδιαλλαγής ήταν το θέμα της χρηματοδότησης των ειδικών μέτρων ασφαλείας, δηλαδή των μέτρων ασφαλείας που δεν είναι τα βασικά μέτρα ασφάλειας τα οποία υπάρχουν σε κάθε αεροδρόμιο, αλλά ε, σε αυτά τα ε, πιο βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα μέτρα τέλο πάντων, τα οποία είναι και πολύ πιο δύσκολο να τα εφαρμόσει κανεί. Μπορώ να θυμηθώ τι συμφωνήσαμε για να μπορέσουμε να εγκρίνουμε την οδηγία. Ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει πράγματι μία πρόταση όσον αφορά τη χρηματοδότηση τη ε, ασφάλεια αεροπορία, λαμβάνοντα υπόψη την άποψη του Κοινοβουλίου, όπω αυτή είχε εκφραστεί στη διαδικασία τη συνδιαλλαγή. Και νομίζω ότι είχαμε συμφωνήσει από αυτού. Τώρα, αυτό τώρα που βλέπουμε σε σχέση με την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι κάτι το πρόχειρο. Δεν αντιμετωπίζει αυτά τα ζητήματα τα οποία είχε θέσει το Κοινοβούλιο στη διαδικασία συνδιαλλαγής ε, και αυτό γιατί το Συμβούλιο κατά πάσα πιθανότητα δεν μπορεί να δεχθεί αυτά που ζητά το Κοινοβούλιο ή γιατί προσπαθούν να βρουν κάποια μέση οδό που δεν είναι αποδεκτή ούτε για τον έναν ούτε για τον άλλον. Δεν ξέρω τέλος πάντων που θα καταλήξουμε ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει θα γίνει ένα κόψε-ράψε των ε, προτάσεων που κανέναν δεν θα ικανοποιήσει. Πού πηγαίνουμε τώρα. Να επανέλθω σε αυτό που είπα προηγουμένως, που ήταν το θέμα των ειδικών μέτρων ασφαλείας. Αν δει κανεί τα πράγματα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, υπάρχουν διάφορε μέθοδοι στα διαφορετικά κράτη-μέλη. Και αυτό το οποίο συμβαίνει τελικά αν θέλουμε να μιλήσουμε σε όρου ε, ενιαίας αγορά, είναι στρέβλωση του ανταγωνισμού γιατί ένα ευρώ πληρώνει κανείς σε ένα αεροδρόμιο για τα τέλη ασφαλείας και στο Ηνωμένο Βασίλειο το άλλο άκρο μπορεί να πληρώσει κανείς 50-60 παραπάνω ευρώ ε, συμβολή στην ασφάλεια. Αυτό βέβαια στρεβλώνει την τιμή του εισιτηρίου και δεν συνιστά ε, δίκαιο ανταγωνισμό εντό ευρωπαϊκή Ένωση. Αν βγει κανεί ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δει για παράδειγμα στι Ηνωμένε Πολιτείε τι γίνεται, η κυβέρνηση εκεί αναλαμβάνει το 100% της, ε, του κόστους ε, για τα αεροδρόμια επί του εδάφους, επί του εδάφους τους. Και μιλάμε για έναν τεράστιο, μια μια τεράστια ε, αγορά, παγκόσμια αγορά. Ε, οι ευρωπαϊκές ε, αεροπορικές εταιρείες ε, και γενικά οι επιβάτες που φεύγουν από αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με όλα τα τέλη που πρέπει να πληρώσουν. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να δω να γίνεται κύριε Πρόεδρε είναι μια λίγο, λίγο διαφορετική πρόταση. Μια πρόταση που αναγνωρίζει ότι ε, θα υπάρχουν ε, διάφορα επίπεδα απειλών σε διάφορα αεροδρόμια, σε διαφορετικά κράτη-μέλη και ότι όλα αυτά τα βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν τα ε, αεροδρόμια σε σχέση με τα διάφορα επίπεδα απειλών αναλαμβάνονται όχι από τον ιδιώτη, τον επιβάτη, αλλά από, σε κρατικό επίπεδο. Πρέπει να υπάρχει γενικώ ένα ε, επίπεδο ασφαλείας στα αεροδρόμια ε, και σε, σε τόπους που είναι προορισμοί ε, επαγγελματικοί. Αλλά κάτι τέτοιο δεν πρέπει να επιβαρύνει τον ιδιώτη επιβάτη. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να πω κάτι, γιατί είναι το τέλος του καταλόγου των ομιλητών. Θα ήθελα να πω κάτι ακόμη σε σχέση με τα ζητήματα που είχαμε συζητήσει στο παρελθόν και ειδικότερα στο ποιος πληρώνει. Θα θυμάστε τη συζήτηση στο παρελθόν που είχαμε και έγινε συνδιαλλαγή και τελικά δεν καταφέραμε τίποτα. Εγώ ήμουν ο μόνος ε, στην αντιπροσωπεία της συνδιαλλαγής που καταψήφισε την συμφωνία ε, που είχα μπροστά. Αντιτάχθηκα στην ομάδα μου ως προς αυτό. Πολλοί είπαν και η κυρία Φώστρη και ο κύριος Αλκαντράου και ο κύριος Μπράτμπουρν. Σωστά ήταν όλα αυτά που είπατε, αλλά το μόνο πράγμα που, είχε που οδήγησε στη συμφωνία αυτή ήταν θα επανέλθουμε ακριβώς σε αυτό το θέμα της χρηματοδότησης, της ασφαλείας. Τότε εγώ δεν ήμουν πολύ ικανοποιημένη, για να σα πω την αλήθεια. Είχα υποπτευθεί ότι αυτό ακριβώ συμβαίνει τώρα θα συνέβαινε. Και βέβαια, Γνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να πληρώσουν τίποτα και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον σημείο όσον αφορά τον, ε, το δίκαιο ανταγωνισμό. Υπάρχει κάποια στρέπλωση γιατί κάποια κράτη-μέλη πληρώνουν, το δικό μου κράτος μέλος ποτέ δεν θα πληρώσει, ανεξαρτήτως του ποιος είναι κυβέρνηση. Ε, ούτως ή άλλως δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, αλλά ε, θα ήθελα να υπενθυμίσω και ότι πρέπει να είμαστε και λίγο ρε, Δεν θέλουμε να στείλουμε τον εισηγητή μας σε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, και ενδεχομένως τη συνδιαλλαγή και να φτάσουμε τελευταία στιγμή να κάνουμε αυτό ε, που κάναμε και την τελευταία φορά, να τον αφήσουμε μόνο του Εάν μου πείτε ότι η χρηματοδότηση της ασφάλειας είναι ένα σημαντικό θέμα και αν μου λέτε ως ε, Επιτροπή ότι είναι ένα θέμα για το οποίο τα, κράτη-μέλη πρέπει να χρηματοδοτήσουν ενισχυμένη ασφάλεια και ακούσαμε και από τον κύριο ε, Ελκαντράου, 35% είναι το κόστος. Μας το είπε το γνωρίζουμε και από περιστατικά στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι θέλει κάποιος να ε, μπει με ένα Land Rover ε, μέσα στο αεροδρόμιο της Γλασκόβης. Ε, όλοι θεωρούν ότι δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει ενισχυμένη ασφάλεια. Αντιθέτως πρέπει τα αεροδρόμια μόνα τους να βρουν έναν τρόπο να χρηματοδοτήσουν τέτοιου είδους περιστατικά. Αν μου πείτε ότι κάτι τέτοιο θέλουμε να το κάνουμε όντω θέμα και αν μου πείτε ότι η Ευρωπαϊκή ότι εμείς ως, Ότι Επιτροπή μπορούμε να πούμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει κάποια χρηματοδότηση της ασφάλειας από τα κράτη-μέλη, ευχαρίστως να το κάνουμε, αλλά να μην φτάσουμε στη συνδιαλλαγή και μετά να ε, υποχωρήσουμε. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σαφείς για το τι θέλουμε να κάνει ο εισηγητής. Και αυτό είναι το μόνο πράγμα που ήθελα να πω επί του θέματος. Λοιπόν, Ματιάς, έχεις το λόγο. Ε, δεν ήθελα να λάβω το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Αλλά μετά από αυτά που είπατε, νομίζω ότι ένα πράγμα είναι απόλυτα σαφές. Πράγματι είναι ντεζαβί, κάτι που έχουμε δει ήδη, κάτι μάλλον που έχουμε ακούσει ήδη στο παρελθόν. Ξέρουμε ότι κανένα κράτος μέλος δεν θέλει να υπομειστεί το σύνολο του κόστους. Κανένας δεν θέλει να πει ότι εμείς θα πούμε να πληρωθεί αυτό από τα κράτη-μέλη και επομένως το Συμβούλιο έχει αυτή την στάση ότι δεν θέλει να ακούσει από την πλευρά του Κοινοβουλίου να πει ότι θα πρέπει να πληρωθεί από τα κράτη-μέλη. Επομένω, ή θα σταθμίσουμε μια γραμμή, θα την κρατήσουμε ό,τι και να συμβεί, ή θα πούμε ότι το θέμα της χρηματοδότησης θα πρέπει να αποκλειστεί από τη διαπραγμάτευση και να προσπαθήσουμε να βρούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα το θέμα να βρούμε μια λύση με το Συμβούλιο. Για μένα το θέμα της χρηματοδότησης είναι δευτερεύον. Προφανώς θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε κάποια στιγμή. Αλλά να είναι σαφές και για το Συμβούλιο τι θέλουμε. Αλλά θα πρέπει να επανέλθουμε κάποια στιγμή για το θέμα αυτό. Και εγώ πιστεύω προσωπικά ότι δεν πρέπει να υποχωρήσουμε ανεξάρτητα από τη θέση του Συμβουλίου να συζητήσουμε τη χρηματοδότηση και να είμαστε συνεκτικοί με αυτό το οποίο έχουμε υποστηρίξει πάντα. Και νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε ως Επιτροπή Μεταφορών εδώ πέρα μια ευρεία συνένεση ότι η ασφάλεια <clears throat> και συγκεκριμένα τα πρόσθετα μέτρα ασφαλείας θα πρέπει να είναι πάντα υπόθεση του κράτους και όχι των καταναλωτών. Αν θέλει λοιπόν κανείς <clears throat> να έχει μια διαφάνεια για τα θέματα αυτά, θα πρέπει να πει ότι αυτό το οποίο εμεί ονομάζουμε πρωτογενή ασφάλεια, ότι το θέμα αυτό θα πρέπει <clears throat> να μην υπόκειται σε τέλη, θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα το καλύπτει το κράτος. Και τώρα, για τα θέματα αυτά, τα θέματα τα οποία ο καταναλωτής δηλαδή πληρώνει το βασικό τέλος, αλλά ό,τι είναι πρόσθετο κόστος, παραδείγματος χάρη κόστος κατά τρομοκρατικής ενέργειας, αυτό θα πρέπει, όπως είπε ο Μπράντμπερν, να το καλύπτει το κράτος. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η άποψη μπορεί να γίνει δεκτή από το Κοινοβούλιο και μας μένει μονάχα το θέμα του αν εμείς θα κρατήσουμε το θέμα αυτό της ε, χρηματοδότησης ή όχι. Αλλά θα πρέπει να έχουμε μια συνακτική θέση για το θέμα αυτό. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω και έχει απόλυτο δίκιο είναι ότι πρέπει να δώσουμε μια κατεύθυνση στον εισηγητή μα για το πού θέλει να πάει. Θέλουμε να συμπεριληφθεί η χρηματοδότηση στην έκθεση. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Με τη μία την άλλη προσέγγιση, κάθε θα κάνουμε. Έχει δίκιο, ό,τι και να αποφασίσουμε. Εμεί, σαν αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου, επιμείνουμε στη θέση μα. Να μην αλλάξουμε κάθε φορά που μυριζόμαστε ότι η ατμόσφαιρα μυρίζει μπαρούτι με το Συμβούλιο και να υποχωρούμε. Αυτό λέω. Πρέπει να υποστηρίξουμε τον εισηγητή ανεξάρτητα από την απόφαση Επιτροπής. Κύριε Κούν, θέλατε σύντομα να πείτε κάτι. Σύντομα και μετά ο κύριο Καγιάκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είδαμε γενικά ότι είναι πεπλεγμένη η κατάσταση. Αυτό φαίνεται από τη συζήτηση και τα πράγματα πράγματι ιστορικά έχουν οδηγήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Μετά το, το μετά από την 11η Σεπτεμβρίου, έχουν οδηγήσει όλα αυτά στο να νιώθει κανείς ότι περισσότερο από οποιαδήποτε μορφή μεταφοράς οι αεροπορικές συγκοινωνίες είναι υπό απειλή και αυτό οδηγεί στα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί. Τώρα, ένας πελάτης ο οποίος αγοράζει ένα αεροπορικό εισιτήριο θα πρέπει να ξέρει ποιο τμήμα του εισιτηρίου, ποιο τμήμα του κόστους έχει να κάνει με την ασφάλεια. Επομένως, το θέμα αυτό της διαφάνειας σε σχέση με τα τέλη ασφαλείας είναι κεφαλαιόδες και το έκανε σαφές και ο εισηγητής. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει και σαφήνεια για όλα τα κράτη-μέλη ποιο είναι το δεσμευτικό επίπεδο ασφαλείας το οποίο πρέπει να εξασφαλιστεί. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει και μια κυριαρχικότητα των κρατών μελών. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να καθορίσουν και να ρυθμίσουν το πώς θα γίνονται οι αστυνομικοί έλεγχοι χάρη των επιβατών στα αεροδρόμια. Και εδώ υπάρχουν διαφορετικές καταστάσεις από το ένα κράτος στο άλλο. Σε ορισμένε περιπτώσεις ήδη έχει γίνει ένα outsourcing, έχει δοθεί σε ιδιωτικούς φορείς αυτός ο έλεγχος ασφαλείας. Σε άλλες παραμένει στα κράτη-μέλη. Είναι σημαντικό να το εξετάσουμε αυτό και υπό την οπτική γωνία της σύγκρισης του κόστους. Αν θέλει λοιπόν η Κομισιόν να εξασφαλίσει ότι υπάρχει συγκριτικότητα σε ό,τι αφορά το κόστος, θα πρέπει να εξετάσει και την πτυχή του ανταγωνισμού. Αν αυτές οι εταιρείε οι οποίες παρέχουν ασφάλεια παραγωγή χάρη, αν παρέχουν το ίδιο επίπεδο ασφάλεια ή αν έχουμε κάτι το οποίο είναι απλώς πολυδάπανο αλλά δεν προσφέρει πρόσφατη, πρόσθετη ασφάλεια. Και επίσης θα πρέπει να είναι υπόλογες αυτές οι εξωτερικές εταιρείες ασφάλειας σε δημόσιους ρυθμιστικούς τομείς. Και θα πρέπει να υπάρχει ο έλεγχός τους από την ε, πολιτική αεροπορία ή από το αεροδρόμιο ανεξάρτητα με την κατάσταση του κράτους μέλους. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει σαφήνεια για το τι καλύπτει το κόστος αυτό και να μην είναι κατά κάποιο τρόπο όλα αυτά τα, αυτές οι πηγές κόστους να είναι ενκρυπτό, να καλύπτονται με άλλο τρόπο. Θα πρέπει λοιπόν μόνο τότε να μπορέσουμε, όταν ξέρουμε ποιο είναι, ποια είναι η πραγματική διάρθρωση του κόστους, μόνο τότε θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια πραγματική ρύθμιση η οποία είναι διάφανη και ισοδίκη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Καγιάκα, κάτι που θέλετε να πείτε, από ό,τι αισθάνομαι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι άκουσε πολύ προσεκτικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έξοχη αυτή συζήτηση και θα ήθελα, όπως και άλλοι ομιλητές, και εγώ να πω στον κύριο Λιχτφριτ, ότι συνόψισε πολύ καλά τα βασικά θέματα. Είπα το ίδιος Πρόεδρε και άλλοι αγορητές το ανέφεραν πως αφετηρία η αφετηρία, η απαρχή του θέματος έχει την όψη déjà vu. Είναι κάτι που ήδη έχουμε δει. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου, όπως εξήγησε η κυρία Φώστερ, ο κύριος Σασάντα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπρεπε να υποβάλει προτάσεις, ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασχοληθεί με την ασφάλεια των ε, αεροδρομίων και της αεροπλοείας και υπάρχει ένα πλαίσιο για το θέμα αυτό στην Ευρώπη. Έγινε μια συζήτηση για καθοριστεί το πλαίσιο που προσφέρει την ευθύνη όσον αφορά την ασφάλεια των αερομεταφορών και κατ' επέκταση που θα πρέπει να πληρώσει για τα σχετικά, οι σχετικές δαπάνες. Οι εμπορευόμενοι, οι κυβερνήσεις ή και οι δύο. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία υιοθετήθηκε τον Μάιο, προσπαθεί να κάνει ένα βήμα παραπάνω και προσπαθεί αυτή την συζήτηση να μετατρέψει σε μια απτή πολιτική. Όμως θα πρέπει να πω ότι η επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του κολεγίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του σώμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν μια ρεαλιστική προσέγγιση. Η πρόταση ακολουθεί μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Φεβρουαρίου που συμπεραίνει ότι μη διακριτικά τέλη και που συνδέονται με, την, με το κόστος ασφάλειας χρειάζονται για να υπάρχει δίκαιο ανταγωνισμό ε, χωρί τρέβλωση μεταξύ αεροπορικών εταιριών και αεροδρομίων. Εκεί που απαιτούνται τέλη, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, θα πρέπει να υπάρχει σχετισμό με το κόστο, να μην υπάρχει διάκριση και θα πρέπει να υπάρξει και διαβούλευση κατά τον καθορισμό των τελών ασφαλείας. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι κάποιε θεμελιώδει αρχέ που δεν γίνονται σεβαστέ τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γίνουν σεβαστέ. Αυτό δεν είναι κάτι μινιμαλιστικό ως προσέγγιση. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τα τέλη αυτά ασφαλείας δεν δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ πληματών και αεροπορικών εταιριών. Πρέπει να εξασφαλίζουμε διαφάνεια και διαβούλευση. Ο κ. Σασάντα κάνει μια ερώτηση. Πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να εξασφαλίσει τη διαφάνεια. Η διαφάνεια μπορεί να εξασφαλιστεί σε τρία επίπεδα ξεχωριστά. Πρώτα απ' όλα σε επίπεδο αεροδρομίων. Οι αεροπορικέ εταιρείε θα πρέπει να παίρνουν πληροφορίε από τα αεροδρόμια όσον αφορά τους φορείς εκείνους που καθορίζουν τις συνιστώσεις μάλλον του κόστους της ασφαλείας σε επίπεδο αεροπορικών εταιριών θα πρέπει οι αεροπορικές εταιρείες να αποφασίζουν ποιες θα πρέπει να είναι οι μελλοντικές επενδύσεις, θα πρέπει να λένε ποιες είναι οι ανάγκες τους οι αεροπορικές εταιρείες και σε επίπεδο κρατών μελών τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι διαφανή όσον αφορά την οικονομική, τον οικονομικό αντίκτυπο των εθνικών μέτρων ασφαλείας που είναι πιο αυστηρά από ό,τι επαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητάμε από τα κάτι μελη να εξετάσουν τον αντίκτυπο των πιο αυστηρών μέτρων που ξεπερνούν τι προδιαγραφέ τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και όπω είπε και η κυρία Φώστερ, και πολύ σωστά το είπε, επίση ζητάμε από τι εθνικέ αρχέ να καθορίσουν ανεξάρτητο φορέα εποπτικό που θα ελέγχει την εκτέλεση της οδηγίας και να διατητεύει όταν υπάρχουν διαφωνήσεις όσον αφορά τα τέλη ασφαλεία. Είπα ότι είναι πραγματιστική αυτή η προσέγγιση. Μια επιλογή πολιτική έγινε. Είπαμε δεν μπορούμε να εναρμονίσουμε τη χρηματοδότηση των τελών ασφαλεία όλη την Ευρώπη. Είναι ανέφικτο. Αν δείτε την αξιολόγηση αντικτύπου θα δείτε τι γίνεται και στα 27 κράτη-μέλη. Η κατάσταση επικύλει σε άλλου τομεί, σε άλλε περιοχές του κόσμου και σε σχέση με άλλε περιοχέ του κόσμου και τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Δεν θα ήταν ρεαλιστική με τέτοια προσέγγιση και ξέρουμε τι έγινε με την οδηγία για τα, τέλη αεροδρομίων. Απέτυχε δύο φορέ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη τρίτη φορά τα καταφέραμε. Ξεκινήσαμε κάνοντα το πρώτο βήμα, επιβάλαμε κάποιε αρχέ, αλλά δεν αγνοούμε το κόστο. Εισάγουμε την αρχή του συσχετισμού με το κόστο. Τα τέλη ασφαλεία θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να καλυφθεί το κόστο ασφαλείας και θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τι χορηγίε και επιδοτήσει που επιτρέπουν οι αρχέ για σκοπού ασφαλείας. Το κόστο των μέσων χρηματοδοτήσεως και το κόστο των εγκαταστάσεων. Υπάρχει συσχετισμό με το κόστο και αυτό μα επιτρέπει να επισέλθουμε στο θέμα. Βεβαίω είναι δικαίωμα του Κοινοβουλίου στην ε, συνδιαλλαγή να πει θα θέλαμε περισσότερα. Θα θέλαμε λιγότερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατανοεί και υποστηρίζει κάποιες ιδέες. Έγινε σημαντική πρόταση. Τα κράτη-μέλη ίσως θα έπρεπε να θεσπίσουν νέα μέτρα, να εφαρμόσουν νέα μέτρα που θα χρηματοδοτούνται για την ασφάλεια. Αυτό είναι ένα θέμα προς συζήτηση. Ακούστηκαν και πλέον φιλόδοξες προτάσεις. Ίσως θα ήταν δυνατόν να υπάρχει ένα αρμονισμένο σύστημα, μεικτό σύστημα, Νομίζω ότι θα είναι δυσκολότατο κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το θέμα της συνδιαλλαγής όμως. Υπήρξαν και θέματα που ετέθησαν για κρατική βοήθεια. Η κυρία Χάνες Πλανσάρτ ανέφερε το θέμα και την ισοτιμία που θα πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει ισότιμο, ισότιμη αντιμετώπιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να αποφύγουμε στρέβλωση του ανταγωνισμού και θεωρούμε ότι εφαρμόζοντας αυτές τις αρχές θα είναι δυνατόν να βελτιώσουμε σημαντικά την κατάσταση, διότι χρειαζόμαστε περισσότερη διαφάνεια. Πρέπει να γνωρίζουμε ποιο είναι ο προορισμό των πόρων. Χρειάζεται περισσότερη διαβούλευση μεταξύ αεροπορικών εταιριών και πιστεύω ότι η οδηγία είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Καθώς και η θέσπιση των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Όπω είπε σωστά ο κ. Δεγράνδες, είναι μεγάλο θέμα αυτό. Η συζήτηση ξεπερνά αυτή την οδηγία. Κύριε Σίμψον, πιστεύω ότι στο κάτω-κάτω εμεί εκφράζουμε την προθυμία μα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχιστούν οι συζητήσει. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια τη συνδιαλλαγή θέλει γενικότερη συζήτηση, ευρύτερη συζήτηση με τα κράτη-μέλη, αυτό είναι δικαίωμα του Κοινοβουλίου και σωστά το θέσατε. Μπορούμε να συζητήσουμε το ποιο πληρώνει, μπορούμε να προσπαθήσουμε να εναρμονίσουμε το σύστημα των τελών αεροδρομίων. Εμεί αποτύχαμε όχι για τα τέλη ασφαλεία, για τα άλλα τέλη αλλά νομίζω ότι έχει βελτιωθεί σημαντικά το κείμενο. Μάλλον είναι σημαντικέ οι βελτιώσει που προτείνει το κείμενο. Έχουμε για πρώτη φορά ένα μέσο που προτείνει ένα σύστημα για την κάλυψη των τελών ασφαλεία. Έχουμε κοινέ αρχέ για πρώτη φορά. Μη διάκριση, διαφάνεια, διαβούλευση, συσχετισμό με το κόστο Και θα ήταν εσφαλμένο να υποτιμήσουμε την αξία του πρώτου βήματο αυτού που μπορεί να οδηγήσει ακολούθω σε περαιτέρω πρόοδο σε έναν τομέα σημαντικότατο. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι το ότι εκφράζει άποψη το Κοινοβούλιο ότι οι συζητήσεις στο Συμβούλιο έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται επί Σουηδικής Προεδρίας και ας εργαστούμε σκληρά για να βρούμε μια λύση κατά τη διάρκεια της συναπόφασης. Αλλά νομίζω ότι θα πάει στη συνδιαλλαγή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Χάνης Πλασά, θέλετε να ξαναπάρετε το λόγο. Σύντομα όμως. Ναι, μόνο μία πρόταση. Όταν είπατε ότι μπορούμε να το συζητήσουμε το ποιος πληρώνει τι, αλλά είπατε επίση ότι δεν μπορούμε να εναρμονίσουμε κλπ. κλπ. Μας κοροϊδέψατε τότε στην προηγούμενη συνδιαλλαγή, στο, στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Μας είχατε πει ότι θα γίνει μία πρόταση και τώρα μας λέτε ότι όχι. Συγγνώμη, θέλω να εκφράσω την διαφωνία μου και τη δυσαρέσκειά μου. Εγώ πάντως καταψήφισα, σας το λέω. Κύριε Λάιτφριντ, θέλετε να απαντήσετε. Να μας δώσετε και ένα χρονοδιάγραμμα, θα σας ήμασταν ευγνώμονες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την τόσο πλούσια και γεμάτη ιδέες και πληροφορίες συζήτηση που μας βοήθησε πάρα πολύ να μπορέσουμε να βρούμε κάποια κατεύθυνση και ακούσαμε όλες τις απόψεις εσείς με αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι έχουν αποσαφινιστεί τα πράγματα ορισμένοι λένε ότι ο ανταγωνισμός δεν πρέπει να αφορά μονάχα τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, αλλά όρο όλο τον ευρωπαϊκό χώρο για να δώσουμε τη δυνατότητα στα αεροδρόμια μας να συναγωνιστούν σε ευρύτερο επίπεδο. Επίσης, τονίστηκε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα σύστημα διαφανές, το οποίο όμως δεν πρέπει να οδηγήσει σε πρόσθετη γραφειοκρατία, σε πρόσθετο κόστος, ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει στον καταναλωτή και σε αεροπορικές εταιρείες να εξασφαλίσουν <clears throat> την σαφήνεια σε σχέση με το τι ζητούν οι ΜΕ και οι ΔΕ. Νομίζω ότι επίσης έχουμε συμφωνήσει ότι εκεί που τα πράγματα λειτουργούν σωστά δεν πρέπει να τα πειράξουμε, ότι πρέπει μονάχα να επέμβουμε όταν δεν λειτουργεί καλά το σύστημα. Όλα αυτά είναι αυτά τα οποία έγιναν σαφέ, σαφή από τη συζήτηση. Και πιστεύω ότι η Επιτροπή μας θέλει επίσης να συζητήσει και το θέμα των τελών ασφαλείας και συγκεκριμένα για το θέμα ποια τμήματα αυτών των τελών θα πρέπει να καλύπτονται από το κοινωνικό σύνολο και πια μόνο από τους χρήστες. Για μένα λοιπόν αυτό το θέμα είναι και το οδηγό νήμα για την έκθεσή μου και θα προσπαθήσω στο βαθμό του δυνατού όσο το δυνατό ταχύτερα να προχωρήσω προς την κατεύθυνση αυτή του να σας δώσω ένα έγγραφο ώστε να μπορέσουμε να ψηφίσουμε τον Δεκέμβριο. Δεν μπορούμε. Όχι λέει ο πρόεδρος Σίμψον. Ίσως είναι πολύ στενά τα χρονοδιαγράμματα τα οποία θέτετε. Περιμένουμε να καταθέσετε το κείμενο της εκθέσεώς σας τον Ιανουάριο και μετά μπορούμε να δούμε πότε θα είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες και πότε θα ψηφιστεί στην Επιτροπή μας. Αν μπορείτε λοιπόν να μου πείτε ότι θα είναι έτοιμη η έκθεσή σας τον Ιανουάριο, εγώ θα σας πω είσαστε ο τέλειος εισηγητής. Πράγματι, αν κάποιο θα ελέγχει όλα αυτά τα πράγματα, αυτό είναι πολύ καλό. Εγώ πράγματι δεν κοίταξα τα χρονοδιαγράμματα. Υπάρχει ένα θέμα ουσίας πάντως, ένα θέμα αρχής, το οποίο θέλω να θέσω ήδη τώρα κλείνοντας. Εγώ προφανώς είμαι έτοιμος για τα θέματα αυτά τα οποία θα φασίσουμε εμείς ως Επιτροπή να βγω στον αγώνα και να παλέψω με το Συμβούλιο. Αλλά θα πρέπει να είμαστε στεναροί για τα θέματα αυτά που θα φασίσουμε και να μην υπαναχωρήσουμε, Αλλιώς δεν έχει νόημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αν έχεις το σχέδιο έκθεσης έτοιμο το Δεκέμβριο, τόσο το καλύτερο. Δεκέμβριο Ιανουάριο είναι πολύ καλά. Και μετά θα δούμε ποια θα είναι η προθεσμία για τις ε, τροπολογίες κλπ. Χρήσιμη η συζήτηση, παρόλο που το έχουμε ξαναδεί, το έργο. Εν πάση περιπτώσει, περνάμε στο επόμενο θέμα της σημερινής διάταξης, που είναι η ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή, ο κύριος Κάχ είναι πάλι εδώ, για το θέμα της κατάργησης των ε, υγρών, για τη μεταφορά υγρών. Σήμερα το πρωί, κύριε Καέκα, ε, συμφωνήσαμε εμείς ε, Φαντάζομαι ότι το γνωρίζετε. Το συζητήσαμε και στους συντονιστές σήμερα το πρωί. Το αποφασίσαμε. Νομίζω λοιπόν ότι ήταν ε, σημαντικό ολόκληρη η Επιτροπή να έχει τη δυνατότητα να ακούσει τι έχει να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, η Επιτροπή σε σχέση με το θέμα της μεταφοράς των υγρών Να δώσω λοιπόν τη δυνατότητα στα μέλη της Επιτροπής να ενημερωθούν καταρχάς και κατά δεύτερον ε, να μας πούν και ιδέες που ενδεχομένως να έχουν δεδομένης ε, της ε, τις θέσεις στην οποία καταλήξαμε. Επίσης καλέσαμε και μέλη της Επιτροπής Ελευθεριών του Πολίτη να έρθουν, να είναι εδώ μαζί μας σήμερα και αν θέλουν να σχολιάσουν και εκείνοι. Η ανταλλαγή απόψεων όμως δεν θα έχει ως αποτέλεσμα κάτι συγκεκριμένο, γιατί την απόφαση την έχουμε ήδη λάβει, αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα θα δώσουμε τη δυνατότητα ε, στα μέλη της Επιτροπής να μας πούν, ε, να μας θέσουν σημαντικά ζητήματα, σημαντικές πτυχές της, ε, του ζητήματος και ενδεχομένως να ακούσουμε και το Συμβούλιο. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι είναι θέμα επιτροπολογίας να σας το υπενθυμίσω αυτό, από ουσιαστικά περιμένουμε τους εμπειρογνώμονες ε, ε, και την υποβολή πρότασης υπό τη διαδικασία της επιτροπολογίας και εμείς μετά λέμε ναι ή όχι απλώς. Δεν μπορούμε τίποτε να τροποποιήσουμε. Ναι ή όχι. Και γι' αυτό θεωρήσα ότι είναι σημαντικό και να καταλήξουμε εμείς σε μια θέση, αλλά να έχουν τη δυνατότητα και τα μέλη της Επιτροπής να ακούσουν πολλά πράγματα για το θέμα. Οπότε, κύριε Καϊκάς. Thank you very much, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαιρετίζει η Κομισιόν την ευκαιρία αυτή να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή σας για το τόσο ενδιαφέρον και τόσο ευαίσθητο ζήτημα και θα ήθελα να σας πληροφορήσω για την κατάσταση των πραγμάτων σε σχέση με τα υγρά. Σας πενθυμίζω εν συντομία τα κύρια στοιχεία της κατάστασης μετά από τα γεγονότα του Αυγούστου 2006 εισήχθη αυτή η απαγόρευση μεταφοράς υγρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από τις <clears throat> τρομοκρατικές απόπειρες που έγιναν ή μάλλον στο Χίθρο. Έχουμε τις πληροφορίες από τις αρχές τις αστυνομικές ότι υπήρχε πράγματι μια σοβαρή απειλή από τα υγρά αυτά και η απαγόρευση εισήχθη ως ένα μέτρο το οποίο θα πρέπει να ισχύει μέχρι ότου η τεχνολογία, η εξέλιξη τεχνολογίας επιτρέπει την άρση αυτού του μέτρου. Ο κανονισμός 272 του 2009 αναφέρει ότι ο κανονισμός αυτός θα εκπνεύσει στις 29 Απριλίου του 2010 με την ελπίδα πάντα ότι θα έχουμε την απαραίτητη τεχνολογία τότε. Πρέπει να σας αναφέρω ότι δυστυχώς οι τεχνολογικές εξελίξεις ήταν πιο βραδίες από ό,τι αναμέναμε και ότι τώρα βρισκόμαστε μόνο σε 7 μήνες πριν από την καθαληφτική ημερομηνία, υπάρχει ένας περιορισμένος αριθμός νέων τεχνικών που είναι διαθέσιμες, αλλά είναι πολύ δύσκολο να έχουν αναπτυχθεί σε όλα τα αεροδρόμια αυτές οι τεχνικές μέχρι τον Απρίλιο του 2010, γιατί τα κράτη-μέλη δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τη διαδικασία προμήθειας αυτών των συστημάτων. Αυτή είναι μια κατάσταση λοιπόν, που πρέπει να αντιμετωπιστεί, όπως είπε και ο Πρόεδρος σας μέσω της Επιτροπολογίας, γι' αυτό ο κύριος Ταγιάννη θέλει να πληροφορήσει στο Κοινοβούλιο σχετικά. Την 1η Οκτωβρίου απέστειλε μια επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών και στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών, πληροφορώντας τους για τα θέματα αυτά. Αν εκπνεύσει αυτή η ρύθμιση που υπάρχει και δεν έχουμε μια εναλλακτική μέθοδο ελέγχου, μπορεί να αντιμετωπίσουμε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί η Κομισιόν έχει πάρει από τις αρχές ασφαλείας πληροφορίες ότι οι απειλές παραμένουν. Δεν υπάρχει άλλη περιοχή στον κόσμο που θα είναι έτοιμη τον Απρίλιο του 2010 για να άρει την απαγορεύση τα υγρά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από την άλλη πλευρά πιστεύει η Κομισιόν ότι θα ήταν λαθασμένο να έχουμε μία παράταση στο διηνεκές των τωρινών ρυθμίσεων. Αν παρατείνουμε χωρίς κάποια ημερομηνία τη συγκεκριμένη <clears throat> ρύθμιση, υπάρχει ο κίνδυνος να διαιωνίσουμε αυτή τη ρύθμιση. Αυτό είναι το χειρότερο που να κάνουμε. Δεν θα στέλνουμε ένα μήνυμα προς τους απαραίτητους κύκλους να, να επιταχύνουν τη δημιουργία συστημάτων ελέγχου. Θέλουμε, επομένως, να επιτρέψουμε να υπάρχουν κάποια υγρά τα οποία θα υπόκεινται σε έλεγχο εν καιρό. Αυτό μπορεί να γίνει μονάχα όμως με ένα σταδιακό τρόπο γιατί δεν μπορούμε όλα τα αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό. Η Κομισιόν λοιπόν θα προτείνει μια σταδιακή προσέγγιση η οποία περιλαμβάνει τρία στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, <clears throat> σαν πρώτο στοιχείο, από το 2010 και μετά τα υγρά, τα εωρήματα και τα αεροσόλ τα οποία προέρχονται από αεροδρόμια εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιτρέπονται σε περιοχές ε, περιορισμένης ασφαλείας και στα αεροπλάνα κάτω από ορισμένε προϋποθέσεις. Αν, είναι, αν υπάρχει απόδειξη ότι έχουν αγοραστεί σε καταστήματα αφορολόγητα και βρίσκονται σε συσκευασία η οποία δεν μπορεί να παραβιαστεί. Δεύτερον, μέχρι τις 29 Απριλίου του 2010, όλα τα αεροδρόμια τα οποία χειρίζονται, από τα οποία διέρχονται μάλλον τουλάχιστον 10 εκατομμύρια επιβάτες κάθε χρόνο, θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να ελέγχουν τα αεροσόλ, τα αερορήματα και τα υγρά όπως προβλέπει ο κανονισμός. Τέλος, μέχρι τις 29 Απριλίου 2010 θα πρέπει σταδιακά μετά από αυτήν την ημερομηνία να εφαρμοστεί αυτή η διαδικασία. Αυτό στην περίπτωση αεροδρομίων που δεν θα είναι έτοιμα και τα οποία θα χρειαστούν πρόσθετο χρόνο. Όλα αυτά όμως θα είναι καταληκτικές ημερομηνίες στα αεροδρόμια, θα πρέπει να μπορούν να ενθαρρυνθούν να το πράξουν αυτό ταχύτερα. Σας τονίζουμε και πάλι ότι αυτή είναι μια πρόταση την οποία θα συζητήσει η Κομισιόν με την Επιτροπή Ασφαλείας της Πολιτικής Αεροπορίας στις 18 Νοεμβρίου. Δεν έχει υπάρξει ακόμα έγκριση αυτής της πρότασης αλλά πριν από τη συνάντηση της Επιτροπής Πολιτικής Αεροπορίας θεωρήσαμε ότι θα ήταν χρήσιμο να έχουμε και τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί θεωρούμε ότι <clears throat> η Κομισιόν θα πρέπει να εξηγήσει στην Επιτροπή Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας ποια είναι η άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό θεωρούμε ότι αυτή η ανταλλαγή απόψεων είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Μετά από τη λήψη απόφαση από την Επιτροπή για την Ασφάλεια της, ε, των πτήσεων, Αφού αποφασίσει, το Κοινοβούλιο φυσικά θα έχει πλήρω το χρόνο να σταθμίσει τη θέση του για τα θέματα αυτά. Λοιπόν, σεβόμαστε τις διαδικασίες, αλλά από αυτή την τρέχουσα ανταλλαγή απόψεων προσπαθούμε να έχουμε και τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω σας τονίσω ότι θα είναι δύσκολη αυτή η συζήτηση στην Επιτροπή ασφάλεια των Πτήσεων. Έχουμε ήδη λάβει σχόλια που λένε ότι αυτού του είδους το χρονοδιάγραμμα που έχει αναφέρει η Κομισιόν είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο. Άλλοι ορισμένοι υποστηρίζουν ένα ανοιχτό χρονοδιάγραμμα, άλλοι θέλουν να έχουν περισσότερο χρόνο. Επίσης υπάρχει διεθνής διάσταση για το θέμα αυτό. Η Κομισιόν είναι έτοιμη να εισαγάγει μια ρήτρα αναθεώρησης εάν οι εξελίξεις δείξουν ότι τα πράγματα προχωρούν ταχύτερα σε διεθνές επίπεδο στην περίπτωση αυτή θα είμαστε έτοιμοι να λάβουμε υπόψη μας αυτές τις εξελίξεις. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει κάτι το οποίο θα λειτουργεί όταν εκπνεύσει η τρέχουσα ρύθμιση. Χωρίς ένα μεταβατικό σύστημα θα βρεθούμε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Πρώτα απ' όλα, γιατί θα έχουμε ένα πρόβλημα ασφαλείας, ένα πραγματικό πρόβλημα ασφαλείας. Δεύτερον, γιατί δεν θα έχουμε κοινού κανόνες στην εσωτερική αγορά. Θα καταληθεί η ενότηση της εσωτερικής αγοράς. Δεν θα μπορούμε να έχουμε ένα μονάχα σημείο ελέγχου του, της ασφάλειας με τις τρίτες χώρες και θα υπάρχει και μια πολυμορφία γιατί το κάθε κράτο μπορεί να εισαγάγει δικά του μέτρα. Θα έχουμε πολλαπλότητα και πληθώρα κανόνων με τις προφανείς επιπλοκές για τους ταξιδεύοντες. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να απαντήσουμε τα ερωτήματά σας, θα λάβουμε υπόψη τις απόψεις που θα διατυπώσετε και θέλω να σας τονίσω ότι υπάρχει μεγάλη πρόοδος σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη νέων συστημάτων. Υπάρχουν τέσσερα είδη τεχνολογία στον τομέα αυτό. Η πιο εξελιγμένη τεχνολογία του τύπου Δέλτα θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο, αλλά είναι ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα σε μια σειρά τεχνολογιών που θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε. Μόλον τούτο θα είναι δύσκολο να προχωρήσουμε στα θέματα αυτά δεν θέλουμε να έχουμε κανόνες που να βασίζονται σε μία και μόνο τεχνολογία. Πρέπει να είναι ουδέτερη ρύθμιση σε σχέση με τις τεχνολογίες, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίζει ορισμένε προδιαγραφέ ασφαλεία. Δεν μπορούμε να λάβουμε κινδύνου. Εναπόκειται στου εμπειρογνώμονε να μα πούν πώ. Θα πρέπει να μείνουμε επίση σε επίπεδο συνεκτικό με τι διεθνεί εξελίξει και συζητούμε το θέμα αυτό με του εταίρου μα και ιδίω με του Αμερικανού, αλλά και με άλλε χώρε όπω η Αυστραλία, ο Καναδά, άλλε χώρε οι οποίε έχουν εξετάσει την ε, τροποποίηση αυτών των κανόνων, χρειαζόμαστε και χρόνο προετοιμασίας. Γι' αυτό το λόγο οι έξι μήνες, εφτά μήνες που μας μένουν δεν είναι επαρκείς. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε εγκαίρως τις απόψεις σας και μετά από την εφαρμογή της διαδικασίας επιτροπολογίας προφανώς το Κοινοβούλιο θα έχει την ευκαιρία να δώσει την ε, άποψή του. Δεν είναι θέμα συναπόφασης, αλλά το Κοινοβούλιο μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη διαδικασία για να εκφράσει την άποψή του. Είμαι έτοιμο λοιπόν να ακούσω τις θέσεις των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσω σε οποιοδήποτε ερώτημα. Όλα αυτά θα είναι πολύτιμα για τη συνάντησή μας 18 Νοεμβρίου με τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ελπίζω να έχουν το σωστό κείμενο τώρα τα μέλη. Ε, της πρότασης των ε, συντονιστών ε, επί της οποίας συμφωνήσαμε σήμερα το πρωί. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε λοιπόν ως ε, κείμενο αναφοράς. Δεν μπορούμε να το τροποποιήσουμε όμως. Μπορείτε όμως να πείτε την άποψή σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να τα λάβει υπόψη. Έχω έναν μεγάλο κατάλογο μιλητών. Και θα είμαι πάρα πολύ αυστηρό με το χρόνο. Δύο λεπτά. Έκαστος. Ο κύριος Κέρκοφ από την Επιτροπή Ελευθεριών του Πολίτη θέλει επίση να πάρει το λόγο και σύντομα γιατί πρέπει να φύγει και θα του δώσω τη δυνατότητα γιατί εμείς στην Επιτροπή Μεταφορών είμαστε πάρα πολύ καλοί και ε, ε φερόμαστε πολύ καλά σε όλους τους ε, υπόλοιπους συναδέλφους. Δεν ξέρω αν αυτό είναι αμοιβαίο, αλλά εν πάση με περιπτώσει εμείς προσπαθούμε. Έχετε δύο λεπτά κύριε Κύρκοφ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ βεβαίως ε, κάνω ό,τι μπορώ ώστε να ανταποδώσω αυτά που κάνετε για μας. Είμαι εδώ από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Έχω κάποιες ανησυχίες, οι οποίες θα ήθελα να εκφράσω. Αυτό που μας ενδιαφέρει έχει να κάνει με τους ε, με την σωματική ακαιρεότητα και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των επιβατών που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Τώρα, τι γίνεται με την κατάσταση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Πρώτα απ' όλα μου φαίνεται ότι πάρα πολλοί άνθρωποι ε, επειδή δεν υπάρχει καλή διαδικασία, επειδή δεν έχουμε τεχνολογία, ε, παραβιάζονται τα δικαιώματά τους. Ε, υπάρχουν κάποιοι επιβάτες που δεν θα πρέπει να είναι στην ίδια κατηγορία ε, με κάποιους άλλους. Επίσης, νομίζω ότι οι ραγδαίες είναι εξελίξεις τεχνολογίας, πολύ πιο σύντομα εξελίσσεται από ό,τι φανταζόμαστε. Δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μην αναβαθμίσουμε τα προηγούμενα μας μηχανήματα, αλλά να αγοράσουμε καινούρια και να, να δημιουργούνται λιγότερα προβλήματα στους επιβάτες. Ε, γι' αυτό από την πλευρά της δικής μας Επιτροπής θέλουμε κάπως πιο αποτελεσματικά να αντιμετωπιστεί το ζήτημα σε σχέση με την πρόταση που βλέπουμε μπροστά μας. Πρέπει να γίνει με έναν τρόπο με τον, με τον οποίο θα ελαχιστοποιούμε ε, τις δυσκολίες που δημιουργούνται στους επιβάτες, να γνωρίζουν επίσης τι πρέπει να κάνουν οι επιβάτες όταν ταξιδεύουν και επίσης λίγη κοινή λογική γιατί υποψιαζόμαστε ότι σε πολλά αεροδρόμια ε, δεν ε, χρησιμοποιείται ιδιαίτερα κοινή λογική όσον αφορά την ανάπτυξη μεθόδων που έχουν στη διάθεσή τους. Δεν χρησιμοποιούνται πάντοτε οι τελευταίες, ε, δεν χρησιμοποιείται πάντοτε η πιο προηγμένη τεχνολογία προς διευκόλυνση των επιβατών. Μάλιστα. Τώρα περνάω στους συντονιστές. Πάρα πολύ σύντομα και πάλι, γιατί είχατε τη δυνατότητα να εκφραστείτε επ' αυτού. Ήδη και τους υπόλοιπους θα θέλαμε να ακούσουμε. Ματιάς, έχεις δύο λεπτά. Ε, ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τρία πράγματα είναι σημαντικά για μας για το θέμα αυτό. Πρώτον είναι η ασφάλεια, αλλά και η κατάλυση όλων αυτών των προβλημάτων και των ενοχλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιβάτες και τρίτον δεν πρέπει να περιμένουμε την τεχνολογία όπως περιμένουν στο θέατρο τον κοντό, θα πρέπει με μεγάλη ταχύτητα να τροποποιηθεί η κατάσταση αυτή. Όλα αυτά λοιπόν οι βασικές βάσεις για μας, είναι σημαντική πρόταση και θεωρούμε ότι οι προθεσμίες θα πρέπει να είναι συντομότερες. Είναι καλύτερα να έχουμε 2012-2013 από ότι 2013-2014. Επίσης δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ των ε, αεροδρομίων και θα πρέπει να χρησιμοποιείται η καλύτερη δυνατή τεχνολογία. Αυτό ίσως μπορεί να μπει μέσα στο κείμενο και δεν θέλουμε να έχουμε να αντιμετωπίσουμε τους ε, λομπίστες οι οποίοι λένε ότι το μοντέλο ότι είναι σε πέντε χρόνια είναι καλύτερο από τα άλλα μοντέλα κτλ. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε την καλύτερη δυνατή τεχνολογία και είναι επίσης πριν από στην Κομισιόν σημαντικό να μπορούμε να έχουμε μια κοινή στάση Κομισιόν και Κοινοβουλίου. Δεν θέλουμε να βρεθούμε μετά τις 29 ε, Απριλίου με 27 διαφορετικά είδη ελέγχου, ένα για κάθε κράτος Αυτό θα είναι ακόμα χειρότερο για τους επιβάτες από το σημερινό ε, καθεστώς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε ποτέ δεν ήμουν υπέρμαχος αυτού του είδους ε, των χρονικών ορίων, αλλά τέλος πάντων. Ήμουν υπέρ, ή μάλλον είμαι υπέρ, της προσεγγίσεως που ακολουθήσαμε πριν. Σταμάτησε η επιτροπολογία. Είπαμε πέρσι ότι θα απαλλαγούμε από την απαγόρευση μέχρι του χρόνου. Εγώ δεν ήμουν υπέρ του μέτρου πρέπει να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή μεταβατική περίοδο. Υποστηρίζω την πρόταση που έγινε να διευκολυνθούν τα πράγματα από τον Απρίλιο 2010 για τους επιβάτες transit με τα φορολόγητα είδη που περνάνε μέσα από τα αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πρέπει να τους διευκολύνουμε αν μπορούμε να το κάνουμε για ενδοκινοτικές πτήσεις πρέπει να γίνει αυτό και πρέπει να καθορίσουμε κάποια προθεσμία, ούτω ώστε να οργανωθούν τα αεροδρόμια. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να πιέσουμε τα αεροδρόμια και τα κράτη-μέλη, ούτω ώστε να κάνουν τις αναγκαίες επενδύσεις, ούτω ώστε οι επιβάτες να διευκολυνθούν. Υπάρχουν τώρα καινούργια συστήματα, η τρίτη γενιά των μηχανημάτων σάρωσης, τα C-scanners, και μπορεί να γίνεται και ξεχωριστή σάρωση, όπως γίνεται με τους φορητούς υπολογιστές, θα μπορεί να γίνει στο μέλλον για τα υγρά. Ίσως αυτό να είναι μεγάλη βελτίωση. Μπορεί να πάρει κανείς ένα μπουκάλι νερό μαζί του στο πλάνο. Μηχάνηματα σάρωσης τόσο εξειδικευμένα θα χρειαστούν κάποιο χρόνο, αλλά πρέπει να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον, τι θα κάνουν και στη ΣΥΠΑ το 2011 στη ΣΥΠΑ κάτι θέλουν να κάνουν πάνω σε αυτό. Και πρέπει να μας ε, δώσει κάποια κατεύθυνση. Αυτά έχω να πω. Ευχαριστώ κύριε κυρία Μάισερ για το Άλτε. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό συμφωνούμε. Θέλουμε περισσότερη ασφάλεια. Ξέρουμε ότι ο τωρινός κανονισμός δεν εξασφαλίζει την ασφάλεια. Θα πρέπει να τον καταργήσουμε, αλλά θα πρέπει να είναι δυνατό να τον καταργήσουμε. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μια πραγματιστική και εφικτή λύση για τις αεροπορικές εταιρείε και για τους ε, επιβάτες που να μην έχει ειδικέ ρυθμίσεις να ισχύει για όλους. Εγώ πιστεύω ότι είναι γρήγορη η τεχνολογία. Πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να εξασφαλίσουμε να έχουμε συστήματα τα οποία θα είναι ευέλικτα και θα εξασφαλίζουν ασφάλεια. Δεν θέλουμε να έχουμε τεράστια συστήματα. Νομίζω λοιπόν ότι το σύστημα ΣΕ είναι αυτό το οποίο μπορεί να λειτουργήσει με κάποιες αναβαθμίσεις. Επομένως, <clears throat> νομίζω ότι είναι καλή η πρόταση της Κομισιόν. Είναι απαραίτητο να υπάρξει μια κάποια ελάφρυνση των ε, επιβατών. Δεν έχει νόημα να υπάρχει ένα κατάστημα φορολογήτων ε, ποτών στη Φραγκφούρτη, αλλά να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν οι επιβάτε λόγω αυτή τη ρύθμιση. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει και μια λογική σε όλα αυτά τα θέματα. Σε ό,τι αφορά το σημείο 2, μπορώ να φανταστώ ότι και το σύστημα τύπου ΔΕΛΤΑ θα είναι έτοιμο το 2013, θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε ορισμένα μεγάλα αεροδρόμια, αλλά αυτό δεν πρέπει να εξαρτάται μονάχα από την απόφαση μονάχα μερικών αεροδρομίων. Ένα άλλο σημείο είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίσαμε προηγουμένως. Προφανώς υπάρχει το κόστος των ε, συσκευών αυτών που κοστίζουν περίπου 300 ε, ευρώ η καθεμία. Εδώ θα πρέπει να βρούμε μια λογική λύση, αν θα το πληρώσουν τα αεροδρόμια ή τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Φώστερ έχει το λόγο για την ομάδα της. Ευχαριστώ, Πρόεδρε θα χαλάσω λίγο την ατμόσφαιρα. Από το 2006 με αυτά τα 100 μιλιλίτρα που μπορούμε να πάρουμε τα υγρά μας έχουν πρίξει. Και όποτε ξεμπερδέψουμε όλα αυτά θα χαρούμε όλους ιδιαίτερος. Κυρίως εκείνοι που γενναιόχονται συχνά. Τώρα υπό την άλλη μου ιδιότητα να πω κάτι. Είδα κάτι πολύ ενδιαφέρον στο Υπουργείο Άμυνας στα επιστημονικά εργαστήρια με τον Πρόεδρο και κάποιους άλλους. Πρόσφατα πήγαμε στον Ηνωμένο Βασίλειο και είδαμε τι κάνουν όσον αφορά με τα υγρά εκρηκτικά και τι μπορούν να κάνουν. Δεν μπορώ να σας τρομάξω, αλλά είναι πραγματικός ο κίνδυνος. Και εγώ δούλευα σε αεροπορικές εταιρείες παλιά και δεν τα παίρνω ελαφρά την καρδία αυτά τα θέματα ασφαλείας. Τούτων λεχθέντων δεν καταλαβαίνω πώς θα προχωρήσουμε τόσο γρήγορα. Δεν βλέπω γιατί να πάμε στον τύπο Γ όταν ξέρουμε ότι έρχεται ο τύπος Δ. Η μετακίνηση στον εξοπλισμό τύπου Γ. Όλοι πρέπει να βγάλουν να τα βγάλουν όλα αυτά, να βγάλουν τα πράγματά τους, να σταθούν σε ουρά τελικά θα μπλέξουν οι επιβάτες σε μεγαλύτερες ουρές με αυτό το σύστημα. Όσον αφορά την πρόοδο μέχρι το μετά το 2010, τέλεια αν το πετύχουμε. Θέμα επιμελητίας, οργάνωσης είναι, είναι πώς είναι φτιαγμένα τα αεροδρόμια. Ε, ασφάλεια στις πύλες. Θα είναι πολύ δύσκολος ο διαχωρισμός. Εγώ είμαι αισιόδοξη, πιστέψτε με. Και θέλω να λειτουργήσουν όλα αυτά. Τούτου λεχθέντος δεν μπορούμε να σπρώχνουμε κάτι το οποίο δεν είναι πρακτικό, δεν είναι ασφαλές και να βιαστούμε κιόλα και να φέρουμε σε δύσκολη θέση εκείνους που θέλουμε να βοηθήσουμε, δηλαδή τους επιβάτες, σε όλο τον κόσμο. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Κρίμερ, για τους πράσινους. Συγγνώμη, προηγουμένως έπρεπε να σου το λόγο, τον πέρδεψα λίγο. Δεν πειράζει είναι παράξενη η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Έχουμε ζητήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς ασφάλεια μας δίνουν αυτοί οι έλεγχοι, γιατί εμείς έχουμε σταθεί εναντίον όλων αυτών των ε, ρυθμίσεων. Μπορεί κανείς να αγοράσει πράγματα, πράγματα από το duty free, να αναμίξει υλικά μέσα στο αεροπλάνο, φέρνοντας στοιχεία από 5 ή 6 επιβάτες και όλα αυτά θα είναι νόμιμα γιατί είμαστε κάτω από το όριο των 100 ml, αλλά μπορούν 6 επιβάτες μαζί να φτάσουν κάτι το οποίο έχει την κρίσιμη μάζα. Εμείς λοιπόν όλοι βασιζόμαστε στην ελπίδα ότι κάποτε θα μπορέσει να βρει η βιομηχανία ένα μηχάνημα το οποίο θα ελέγξει τα πάντα. Αλλά ξέρουμε ότι αυτό δεν υπάρχει ακόμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει ένα σφάλμα και αυτή τη στιγμή ετοιμαζόμαστε να συνεχίσουμε αυτό το σφάλμα, να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερη γραφειοκρατία και να πολλαπλασιάσουμε αυτό το σφάλμα. Μιλήσαμε ήδη για το κόστος της χρηματοδότησης, ότι κοστίζουν 300 ευρώ αυτά τα, αυτή, εξώ, αυτά τα, τα μηχανήματα. Με τον τρόπο αυτό δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Εγώ νομίζω ότι το πρώτο βήμα το οποίο κάναμε το να εφαρμόσουμε αυτούς τους καν, κανόνες ασφαλείας ήταν απατηλό, ήταν λαθασμένο. Δεν νομίζω ότι μπορούμε πράγματι να εξασφαλίσουμε τα κριτήρια ασφαλείας τα οποία λέμε ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε ακόμα και στις ημερομηνίες που έχουν προταθεί. Κυρία Βόρτμαν Κόλ. Και πάλι. Δύο λεπτά είναι δυνατόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, θέλω να πω ότι συμφωνώ με αυτό το οποίο είπε ο κύριος Κράμερ προηγουμένως. Έχουμε νιώσει πραγματικά εξοργισμένοι μερικές φορές τα τελευταία χρόνια γιατί κανείς δεν μπορεί να μας εξασφαλίσει ότι υπάρχει μια ασφάλεια. Όταν πέρσι μας λέγανε ότι θα γίνει πραγματικότητα αυτή η ημερομηνία της 29ης Απριλίου 2010 ήμασταν ικανοποιημένοι. Τώρα μας λένε ότι αυτό είναι αδύνατο να γίνει στην πραγματικότητα. Δεν ξέρω λοιπόν ποιος φταίει αυτή τη στιγμή. Και δεν ξέρω αν θα πρέπει να μιλάμε για το 2014, αν πρέπει να μιλάμε για φουτουριστικές τεχνολογίες τύπου Δέλτα και όλα αυτά. Εγώ φοβάμαι ότι με μια τέτοια αναβολή θα καταλήξουμε και πάλι στο να μην υπάρξει καμία κατάργηση. Οι συντονιστές μας είχαν αποδεχθεί να ισχύσει αυτή η ημερομηνία της 29ης του 2010 επί τη βάση της καλύτερης υπάρχουσας τεχνολογίας όπως είπε και ο κύριος Γκρός. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2013 την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία. Επίσης, αυτό ήταν το πρώτο μου σημείο, επίσης είναι γεγονός ότι υπήρξαν πολλά παράπονα για το γεγονός ότι ορισμένα, ε, ορισμένες ουσίες δεν μπορούν να τις μεταφέρουν οι επιβάτες στα αεροδρόμια. Αυτό δημιουργεί πραγματικά πάρα πολλά προβλήματα στα αεροδρόμια και χρειάζεται και λίγη περισσότερη φαντασία για να βρούμε λύσεις σε όλα αυτά τα προβλήματα. Και υπάρχει επίσης και ένα μεγάλο πρόβλημα γιατί ορισμένα αεροδρόμια αντιμετωπίσουν με μεγάλη αυστηρότητα αυτά τα μέτρα, ενώ άλλα είναι πολύ χαλαρά. Αυτό ενοχλεί του επιβάτε. Θα πρέπει να υπάρξει μια μεγαλύτερη ομοιομορφία τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομο γιατί υπόθηκαν ήδη πολλά. Κοιτάξτε, είναι λίγο μάταιη αυτή η συζήτηση, γιατί σήμερα μας λένε πριν από το τέλος της προεδρίας μερικούς, της προθεσμίας, τους τελευταίους ε, μήνες, ότι δεν προλαβαίνουμε και λέμε ότι πρέπει να ζητήσουμε από τους υπεύθυνους, από τους κατασκευαστές ε, να είναι έτοιμη η τεχνολογία ως τότε. Σήμερα ε, μας ζητάτε να πάμε λίγο πιο γρήγορα από αυτό που έχει προβλέψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα επικέστερης ε, ασφάλειας ε, απλώς να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες καταστάσεις στα διάφορα δρόμια όπου υπάρχουν κάποιες δυσλειτουργίες, εν πάση περιπτώσει, λόγω αυτής της κατάστασης. Αλλά αυτό που θα ήθελα να πω, έτσι μια μικρή διαφωνία σε σχέση με αυτό που είπε... Με, με, ως προς την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι σημαντικό να έχουμε μία και μοναδική ημερομηνία εφαρμογής ε, και να υπάρξει και σαφήνεια και διαφάνεια από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής μεγαλύτερη ε, σε σχέση με αυτήν την ε, ισορροπία που πρέπει να εξεύρουμε και με τους κατασκευαστές εφόσον εξαρτάται από αυτούς. Ευχαριστώ πολύ θα ήθελα και εγώ να πω ότι στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία η ομάδα μου δεν συμφωνούσε. Είχαμε πολλές φορές δείξει πόσες, πόσο αναποτελεσματικό ήταν αυτό το μέτρο και ζητήσαμε την κατάργηση πολλές φορές. Ασκήσαμε τις σχετικές πιέσεις ώστε να υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι ελέγχου. Είναι μάλλον ε, εκπληκτικό το γεγονός ε, ότι δεν μπορούμε να σεβαστούμε την προθεσμία της της 9 η Απριλίου του 2010, αλλά πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, και όπως και οι δικοί σας συντονιστές, θα ήθελα να πω ότι ε, δεν θέλουμε να, μεγαλύσουμε, να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη ε, σύγχυση και δεν θέλουμε μια περιπτωσιακή προσέγγιση γιατί θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Εκεί που διαφωνώ είναι Βεβαίω θέλουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση των επιβατών. Το θέμα είναι να το κάνουμε με έναν τρόπο που να είναι εφικτό. Οι αεροπορικές εταιρείε που έχουν ασφάλεια ε, στις ε, ε, πύλες Ε, πολλές φορές δημιουργούν πολύ μεγάλο πρόβλημα στην κίνηση και ίσως ε, πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό. Τώρα όσον αφορά την, ε, την τεχνολογία τύπου C, νομίζω ότι είναι ο, καλ, ο καλύτερος τρόπος. Βέβαια υπάρχει και η τεχνολογία D, είναι η καλύτερη λύση, αλλά δεν την έχουμε ακόμη στη διάθεσή μας. Είπαμε ότι σε 18 μήνες μπορούμε να, το έχουμε, να έχουμε τον τεχνολογικό εξοπλισμό στη διάθεσή μας. Μπορούμε όμως να το κάνουμε. Ε, και αν όχι, τα τύπου ή μηχανήματα είναι καλά για τις ΗΠΑ. Γιατί όχι για μας. Το είπε και ο κύριος Ελκαντράουι προηγουμένως. Ε, αν είναι δυνατόν τα μηχανήματα ελέγχου των υγρών να τα έχουμε το 2011, ε, τότε τι ακριβώς κάνουμε εδώ είτε πρόκειται για τύπου B είτε πρόκειται για τύπου C το θέμα είναι γίνεται αξιολόγηση της ροής των επιβατών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα, στα αεροδρόμια. Νομίζω ότι στη χειρότερη περίπτωση το 2012 θα μπορούσαμε να είχαμε την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Ευχαριστώ. Πάρτε λοιπόν ανάσα, κύριε κυρία για τους πράσινους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα συνεχίσω σε αυτά που είπε η συνάδελφος Κράμερ Νομίζω ότι όταν θα πρέπει να αξιολογήσουμε ένα σύστημα προτού αναπτύξουμε κάποιο άλλο, θα πρέπει να ξαναθέσουμε τα ερωτηματικά. Ο κ. Καράτα ξέρει και, όπως και εγώ ότι το 2001 όταν θεσπίσαμε τον κανόνα όσον αφορά τα αιχμηρά αντικείμενα ήταν υπό την επίρρεια της 11 Σεπτεμβρίου. Η δεύτερη απόφαση όσον αφορά τα υγρά ήταν απόφαση που ελήφθη, έπρεπε να ληφθεί αμέσως μετά τα σοβαρότατα γεγονότα. Αρκετά χρόνια μετά που δεν έχουμε την βέβαιη απόδειξη ότι υπάρχει μια προστασία πραγματική για τις αερομεταφορές και τους επιβάτες, είναι η στιγμή να θέσουμε το ερώτημα. Ε, θα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή δεν είχε η δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποχρεώσει τον τομέα να μεταμορφωθεί. Αυτό είναι το ερώτημα που έχει τεθεί. Θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερωτηθεί για τις επιλογές της όσον αφορά τον αριθμό των λίτρων νερού και σαμπουάν που είναι, αποθηκεύονται ε, στα αεροδρόμια, που κοστίζουν σε χρόνο εργαζόμενους πτήσεις που έχουν χαθεί από όλια σλότια τα αεροπλάνα να δουν πόσο κοστίζουν αυτοί οι έλεγχοι. Και αν πάνε σε σύστημα γ, δ, ε, σ, τ, κλπ. Ε, θα αυξηθεί ο χρόνος ελέγχου κάποιων υγρών. Τώρα εκεί θα πρέπει να διαρωτηθούμε. Τώρα ή ποτέ. Ισορροπία μεταξύ ασφαλεία από τη μία πλευρά και κόστου ή δαπανών. Το σύνολο των δαπανών που αντιπροσωπεύει ένα μέτρο που θα μπορούσε να περιπλέξει την περαιτέρω τον έλεγχο των επιβατών των χειραποσκευών. Να θυμηθούμε ότι υπάρχουν και υγρά εντό τη βαλίτσα και υπάρχει ε, στον αποθηκευτικό χώρο του αεροσκάφου. Μπάμε το έχει στη χειραποσκευή, το έχει στη βαλίτσα. Τώρα ήρθε η στιγμή να γίνει μια πραγματική αξιολόγηση τη σχέση ασφάλεια, δηλαδή ωφέλου πριν προχωρήσουμε προς άλλες προθεσμίες, προς άλλα μέτρα. Ευχαριστώ, κύριε Βαντάλεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι άκουσα προσεκτικά αυτά που υπόθηκαν και αυτά που αποφάσισαν οι συντονιστές. Αλλά όσον αφορά τους ε, επιβάτες που περνούν τράνζιτ, είναι σαφές ότι υπάρχουν τρία μεγάλα αεροδρόμια που θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα Βιέννη, Βερολίνο και Άμστερνταμ. Αυτά τα τρία αεροδρόμια θα έχουν πρόβλημα. Διότι κάνουν ελέγχου στην πύλη και στο χώρο πίσω από αυτόν μπορούν να αναμειχθούν οι επιβάτες τράνζιτ με τους άλλους επιβάτες και θα υπάρξουν τεράστιες ουρές σε αυτά τα αεροδρόμια οπότε μπορούμε εδώ να παίρνουμε γρήγορα αποφάσεις αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε και όλες τις συνέπειες των αποφάσεων. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, κατά πόσο είναι διαθέσιμη τεχνολογία Γ ή όχι. Ο τύπος Δ θα είναι σε δύο χρόνια έτοιμος. Θα πρέπει στο 2 λοιπόν να προσθέσουμε τουλάχιστον τύπου Γ. Τρίτο, Πρόεδρε, ένα ερώτημα προς εσάς. Έχει νόημα αυτή η συζήτηση. Όλοι μπορούμε να συζητάμε μεταξύ μας. Αλλά έτσι που έχουν τα πράγματα με τη συζήτηση όπως πάει, δεν νομίζω ότι θα βγει κάποιο αποτέλεσμα. Ε, δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε κάτι για το κείμενο τελικά. Κύριε Βαντάλεν, δεν μπορεί να κάθεται κανείς σε μια συνεδρίαση και να, σε μια συνεδρίαση να συμφωνείς και σε άλλη συνεδρίαση να διαφωνείς. Ήσασταν σε συνεδρίαση συντονιστών και δεν είπατε τίποτα αντίθετα στο κείμενο ε, που συμφώνησαν οι συντονιστές. Αυτό είναι δικό σας πρόβλημα. Ο κύριος Βαντάλεν, θα ήθελα να πω κάτι πάνω σε αυτό. Εγώ στη δεύτερη ανάγνωση το είπα. Μπορείς να παρεμβαίνει, κύριε Βαντάλεν όταν ε, το επιτρέπει ο πρόεδρος. Θέλετε να παρέμβετε. καλώ, λέει ο πρόεδρος. Όλη αυτή η διαδικασία ίσως θα πρέπει <clears throat> να τις σκεφτούμε υπό την οπτική γωνία ανθρώπων που βρίσκονται σε αεροπλάνα και αεροδρόμια και δεν μπορούν να αποφύγουν όλα αυτά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για αυτούς να ξέρουν τι ακριβώς θα συμβεί. Νομίζω ότι θα πρέπει τουλάχιστον να γίνει δημόσιο αυτό το οποίο αποφασίζουμε. Να μην του πούμε ότι θα ξέρουμε μονάχα σε τρία χρόνια τι θα γίνει. Δεν μπορούμε να περιμένουν και να ανέχονται αυτή την κατάσταση οι πολίτες ακόμα περισσότερα χρόνια. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρξει σωστή πληροφόρηση και σαφήνεια για τους επιβάτες, για τα αεροδρόμια, για τις εταιρείες, να γνωρίζουν τι θα λέει αυτή η νέα ρύθμιση και ότι θα είναι υποχρεωτική. Αυτή τη στιγμή στα αεροδρόμια βλέπει κανείς διαφορετικές ανακοινώσεις οι οποίες ποικίνουν από το ένα αεροδρόμιο στο άλλο και φυσικά υπάρχουν διαφορές και ποικιλία μεταξύ των κρατών μελών. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν αυτή την ομοιομορφία και εμείς τώρα βρισκόμαστε στο τέλος του 2009. Από το 2006 βρισκόμαστε στο 2009. Δεν μπορεί να περιμένουμε άλλα πέντε χρόνια μέχρι να έχουμε τις κατάλληλες συσκευές. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει απαραίτητη πίεση σε αυτούς οι οποίοι αναπτύσσουν αυτά τα μηχανήματα για να κρατήσουν, για να τηρήσουν τα χρονοδιαγραμμάτα που έχουμε πει. Η κυρία Μποσκούρτ έχει τώρα το λόγο. Κυρία Μποσκούρτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι, εγώ είμαι κύριε Πρόεδρε. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Και εγώ έρχομαι από μια άλλη επιτροπή. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που απευθύνατε στα μέλη της Επιτροπής Δημοσίου Ελευθεριών. Θα ήθελα και εγώ να θέσω ένα ερώτημα εδώ. Γιατί αναρωτιέμαι τι ακριβώς λέμε εδώ. Μιλάμε για το συμφέρον των αεροδρομίων, για το συμφέρον των επιβατών, οι οποίοι πράγματι αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Θέλω λοιπόν να σταθώ σε ορισμένα σημεία. Καταρχήν, αυτά τα οποία λέγονται για τα πραγματικά προβλήματα ασφάλειας. Πώς είναι δυνατόν όταν εγώ πετάω από το Παναμά ως το Άμστερνταμ να έρχομαι με δύο μπουκάλια που είναι του μισού λίτρου και να μην με ελέγχει κανένας και μετά να πετάω από το Άμστερνταμ στην Κοπενχάγη και να υπόκειμε σε χιλιάδες ελέγχους. Τα 200 χιλιόμετρα από το Άμστερνταμ στην Κοπεχάγη γίνεται χαμός στους ελέγχους και τα 2.000 από τον Παναμά δεν γίνεται τίποτα. Και επίσης, Βλέπουμε στα αεροδρόμια ότι δεν υπάρχει ακόμα έτοιμη τεχνολογία. Μα λένε οι βιομηχανίε ότι όλα είναι έτοιμα και στι ΗΠΑ τα έχουμε ελέγξει όλα. Αλλά θα ήθελα να ξέρω τι πιστεύει η Κομισιόν σε όλα αυτά τα πράγματα και να μα εξηγήσει ποια είναι η πραγματική κατάσταση. Ο κ. Δεγκράντε Πασκουάλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προσπαθώ και εγώ να είμαι σύντομο όπω μου το ζητήσατε. Εγώ δεν θέλω να, να ξεχάσουμε ένα σημαντικό στοιχείο. Όλε αυτέ οι μορφέ περιορισμού έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των επιβατών από τρομοκρατικές ενέργειες. Είναι πολύ εύκολο να πυροβολεί κανείς την Κομισιόν και να λέει ότι η Κομισιόν είναι ανίκανη. Είναι πολύ εύκολο να κάνουμε λαϊκιστικές κορώνες για τους πολίτες μας και να πούμε ότι η Κομισιόν δεν μπορεί να τα κάνει αυτά τα οποία λέει θα πρέπει να γίνει. Πρέπει να πούμε ότι, ότι μετά από τις 29 Απριλίου του 2010 θα πρέπει να έχουμε ένα πλαίσιο αποφάσεις. Και αυτά μπορούν να γίνουν μονάχα μέσα στα πλαίσια της επιτροπολογίας. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η στάση μας πρέπει να είναι πραγματικά ζυγισμένη και σταθμισμένη. Δεν θα εξαφανιστεί η τρομοκρατική απειλή. Δεν μπορούμε να πούμε στους τρομοκράτες ότι κοιτάξτε, καθυστερήστε λιγάκι, γιατί εμεί δεν μπορούμε να βρούμε μία μέθοδο για να σα αναχαιτήσουμε. Και προφανώ θα πρέπει εμεί να συζητήσουμε σοβαρά με την Κομισιόν για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα σύστημα πριν από τι 29 Απριλίου 2010, το οποίο να είναι σοβαρό και να μην ενοχλεί του πολίτε τόσο πολύ. Αλλά δεν δεν πρέπει να ξεχάσουμε όμω ότι ο αγώνα για την κατάσταση τη τρομοκρατία είναι ο βασικό στόχο μα και δεν μπορούμε εκεί πέρα να κατεβάσουμε τι ασπίδε μα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω Συμφωνώ με τον ε, προαλήσαντα συνάδελφο, αλλά και με άλλους. Ε, βεβαίως θέλουμε να μην υπάρχει δυσκολία και να διευκολυνθούν ε, οι επιβάτες και η ασφάλεια δεν γίνεται ποτέ να παραγωνιστεί. Αλλά αν οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν εγκρίνει τον τύπο C και όποιο πάει στι Ηνωμένε Πολιτείε ή εντό των Ηνωμένων Πολιτειών γνωρίζει ότι εμείς έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο καθεστώς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όποιος λοιπόν πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, θα δει ότι τα συστήματα ασφαλείας είναι πολύ καλύτερα από ό,τι αυτά που έχουμε εμείς εδώ. Νομίζω ότι το τύπος Γ, λοιπόν, τύπος Σ είναι τα μηχανήματα τα οποία θα έπρεπε να ε, έχουμε και εμείς. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι βέβαια ε, θα υπάρχουν και πολύ μεγαλύτερες ουρές και η ροή των επιβατών θα είναι πολύ μικρότερη αλλά έχουμε πολύ συζητήσει το θέμα ε, της ε, ε, εναέριας ασφάλειας και πρέπει κάποτε να το συσχετίσουμε και με την τεχνολογία που έχουμε. Υπάρχει κανένας άλλος που θέλει να πάρει το λόγο? Θα σας δώσω ένα λεπτό, γιατί μιλήσατε και προηγουμένως. Για την ασφάλεια και πάλι. Με τις μεθόδους που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πραγματικά καμία ασφάλεια. Βλέπουμε ότι και ο τύπος σε δεν είναι αρκετά ακριβή στις ΗΠΑ για να μας δώσει ασφάλεια. Και εγώ τόνισα ότι πρέπει να αλλάξουμε το σημείο 2 και να πούμε το 2013 ή όταν έχουμε την κατάλληλη τεχνολογία. Είναι απαραίτητο να λέμε 2013. Αλλά το θέμα είναι αν θα μπορέσουμε να το εξασφαλίσουμε, γιατί πρέπει να έχουμε την κατάλληλη τεχνολογία. Θέλουμε να έχουμε το τύπο Γ, το τύπο Σ ή όχι. Εντάξει, κάποιος άλλος θέλει να πει κάτι. Να προσπαθήσω να κάνω κάτι σαφές σε όλους, γιατί υπάρχει μεγάλη σύγχυση. Εγώ μίλησα με τις εταιρείες που παράγουν τα μηχανήματα. Μια από αυτές τις εταιρείες βρίσκεται στη δική μου εκλογική περιφέρεια και της κυρίας Φώστερ Μίλησα στη Smith που είναι μια από τι μεγάλε αυτέ εταιρείε και οι δύο μου είπαν ανεξάρτητα ο τύπο Δέλτα είναι 5 ή 7 ή 8 χρόνια πίσω από τις άλλες τεχνολογίες. Δεν πρόκειται να είναι έτοιμο, έτοιμα τα μηχανήματα τύπου Δέλτα εγκαίρως. Αυτό μας αφήνει με τον τύπο ΣΕΦ. Δεν είναι ακριβώς έτοιμος ο τύπος ΣΥ, αλλά θεωρούν ότι μέσα στον επόμενο χρόνο θα υπάρχουν μηχανήματα τύπου σε αναβαθμισμένα που θα είναι έτοιμα. Οι Ηνωμένε Πολιτείες χρησιμοποιεί τα αναβαθμισμένα μηχανήματα τύπου σε, επομένως ούτε και οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν μια συγκεκριμένη ημερομηνία για το πότε θα είναι έτοιμα αυτά τα μηχανήματα, παρά το γεγονό ότι δηλώνουν ότι ελπίζουν ότι θα γίνει αυτό το 2011 τύπος Δέλτα που να είναι έτοιμος και να γυαλίζει και να λειτουργεί τέλεια, θέλουμε 8 με 10 χρόνια. Ο τύπος C αναβαθμισμένος μπορεί να είναι πραγματικότητα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια και αυτό κάνουν προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι Αμερικανοί. Θα πρέπει λοιπόν να καταλαβαίνετε ποια είναι η κατάσταση. Γι' αυτό έχει αυτή τη διατύπωση η δεύτερη παράγραφος γιατί πρέπει να εξασφαλίσουμε τη διαδικασία πιστοποίησης σε όλα τα κράτη-μέλη προτού να χρησιμοποιηθούν αυτά τα μηχανήματα. Αυτό σημαίνει επίσης ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ό,τι άλλη διαθέσιμη τεχνολογία υπάρχει εάν υπάρξει μια νέα τεχνολογία για να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα. Απλώς θέλω λοιπόν να σας εξασφαλίσω ότι θα έχετε συνειδητοποιηθεί για αυτό το θέμα. Γι' αυτό οι συντονιστέ καταλήξαν σε αυτή τη θέση. Με μια μακρά συζήτηση με την παρουσία του κ. Καλιάκ, καταλήξαμε σε αυτή την θέση. Είναι διαφορετική από τη θέση κίνησής μα γιατί έτσι μας έφεραν τα πράγματα. Τώρα, σε σχέση με, την, το ρόλο του Κοινοβουλίου στη λήψη αποφάσεων, δεν έχουμε ένα ρόλο για την διαμόρφωση των αποφάσεων σε αυτή τη φάση. Ο ρόλος μας είναι να πούμε ναι ή όχι στο τι θα πούν οι εμπειρογνώμονες και οι κομισιόν μέσα στη διαδικασία της επιτροπολογίας. Αυτό που προσπαθώ εγώ να κάνω είναι να σας δώσω μια ευκαιρία να ακουστεί η φωνή σας βασικά, παρά το γεγονός ότι μερικοί από εσάς θεωρούν ότι αυτό είναι απώλεια χρόνου. Εγώ θα μπορούσα να πω από την αρχή αυτό το θέμα είναι θέμα επιτροπολογίας και πρέπει να το συζητήσουμε μονάχα βάσει της διαδικασίας επιτροπολογίας αλλά πιστεύω ότι θέλετε να εκφράσετε τις απόψεις σας και επίσης έπρεπε και οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Δημοσίου Ελευθεριών να έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν την γνώμη τους. Η πρόταση λοιπόν την οποία εμεί έχουμε διατυπώσει είναι μια απάντηση στην πρόταση της Κομισιόν που όλοι συμφωνούν ότι δεν είναι ο τρόπος να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Εάν πρόκειται να πούμε στην Κομισιόν δεν είναι αυτή η λύση που μας προτείνεται, θα πρέπει να έχουμε και κάτι το οποίο θα παρουσιάσουμε από την πλευρά του Κοινοβουλίου να του πούμε λειτουργήστε με αυτή τη βάση σε τελική ανάλυση, αν θέλουν να το αγνοήσουν, ούσο τους καπέλο τους. Εάν αυτή είναι η απόφαση των εμπειρογνωμόνων, πάλι δικό τους θέμα. Εμείς τελικά θα πρέπει να αποφασίσουμε να δεχτούμε ή να απορρίψουμε την τελική θέση της Κομισιόν. Αλλά οι εξουσίες του Κοινοβουλίου δεν θα ασκηθούν σε αυτό το επίπεδο, θα ασκηθούν στο επόμενο στάδιο. Απλώς μας δόθηκε η ευκαιρία να έχουμε μια πλήρη συζήτηση με την παρουσία της Κομισιόν, η οποία μπορεί να μεταφέρει το μήνυμά σας στην Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων. 30 δευτερόλεπτα. Ναι, ναι, είσαστε ο πρόεδρος. Ευχαριστούμε που έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε. Είμαι μέλος και αυτής της Επιτροπής και της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών. Αλλά το ερώτημα το οποίο έθεσα σε εσά σε σχέση με την απόφαση των συντονιστών για τους μετεπιβαζόμενους ε, επιβάτες, γιατί αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα για ορισμένα αεροδρόμια. Ένα αεροδρόμιο, το Σίπχολ, αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα οργανωτικά, διότι έχουν υιοθετήσει μια διαδικασία ελέγχου στις πύλες. Αν δείτε το μέγεθος των ροών, Βιέννη, Βερολίνο, Χήθρο, Σίπχολ, αν κάνετε σύγκριση, το πρόβλημα είναι το Σίπχολ. Ένας από τους λόγους τους οποίους είμαι αντίθετος και λέω ότι δεν θέλω να πούμε να το έχουμε έτοιμο το 2011, διότι πρώτα απ' όλα πρέπει να αναπτυχθεί η τεχνολογία, αλλά πρέπει να επιτρέψουμε και στα προβληματικά αεροδρόμια να προσπαθήσουν να προσαρμοστούν. Δεν θέλω να επιτεθώ κατά του ΣΥΠΟΛ. Δεν είναι ένα θέμα που φορά μέσα του ΣΥΠΟΛ ένα από τα προβλήματα, είμαστε ειλικρινεί, είναι ότι πέρσι ξόδεψαν πολλά χρήματα στα μηχανήματα και δεν θέλουν να ξοδέψουν και άλλα χρήματα σε τρία χρόνια. Και πρέπει να προσέξουμε τα αεροδρόμια, διότι πολλά αεροδρόμια που διαμαρτυρήθηκαν, δεν διαμαρτυρήθηκαν θέματα ασφαλεία, όπω είπε και ο κ. Γκάντε Πασκουάλ, δεν θέλουν να δώσουν χρήματα διότι θεωρούν ότι αυτό θα του συμβεί. Θέλουν να το δούμε σαν θέμα ασφαλεία, όχι τι γίνεται με το Μάντσεστερ, το Σιπχολ, πρέπει να είναι ένα κομμάτι της γενικής εξέτασης από των τεχνικών ειδικών και ίσως μας πούν αυτό δεν λειτουργεί για τον τάδε ή λόγο. Δεν θέλω να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες προβλημάτων συγκεκριμένων ευδομίων. Είναι ένα πρόβλημα όταν γίνεται ο έλεγχος της πύλης και όχι γενικός έλεγχος. είναι περισσότερο πρόβλημα στις Ηνωμένε Πολιτείε και δεν θεωρούν θα υπάρξει πρόβλημα όταν εισαχθεί το αναβαθμισμένο μηχάνημα τύπου C. Διάλογος εκτός μικροφώνου. Απάντηση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχαμε, κυρίως όσον αφορά από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, είναι ότι τους έκλεβαν, έκλεβαν τους επιβάτες τα duty free. Δεν μπορεί να έχει και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Προσπαθούμε. Οι επιβάτες transit με τα φορολόγητα να περνάνε πιο γρήγορα διαχωρίζοντάς τους. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα πρόβλημα οργανωτικό. Όμως, στο τέλος, στο κάτω-κάτω, εμείς θέλουμε να θέσουμε τέρμα να λυθεί το πρόβλημα εκείνων που έχουν αγοράσει νόμιμα αγαθά και τους αφαιρούνται. Γιατί έχουν να πετάξουν άλλα 100 μίλια εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και γι' αυτό έχουμε την πρώτη παράγραφο. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα με τους επιβάτες που περνάνε, που είναι σε τράνζιτ. Αυτές είναι απλές προτάσεις. Δεν έχουμε καμία εξουσία να τα επιβάλλουμε αυτά. Καλώς το ξέρα θα συνέβαινε αυτό. Η κυρία Λότφορντ έχει το λόγο. Λυπάμαι, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, είμαστε σίγουροι, είσαστε σίγουρος ότι τα οργανωτικά προβλήματα διαχωρισμού των επιβατών τράνζιτα τους άλλους δεν δημιουργούν κενά ασφαλείας αν υπάρχει διαφορετική ε, μεταχείριση των μεταβιβαζομένων επιβατών από τους άλλους. Μετεπιβιβαζομένων μάλλον επιβατών. Εγώ δεν είμαι σίγουρος για τίποτα, δεν είμαι ειδικό για τα θέματα ασφαλείας, λέει ο Πρόεδρος. Θέλω να δω θα που είναι ειδικοί σε σχέση με αυτά που λέμε. Εμείς τους ζητάμε να εξετάσουν το θέμα των επιβατών transit από τους οποίους κατάσχονται τα υγρά διότι θεωρούμε ότι αυτή είναι νομιμοποιημένη κλοπή. Και αυτό τους ζητάμε να εξετάσουν. κυρία Βότμαν Κόλ. Συγγνώμη, αυτή η συζήτηση 30 δευτερόλεπτα δώσατε και δεν θα πρέπει να μπούμε στι τεχνικέ λεπτομέρειε. Αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε και όταν θα ακούσουμε του επιρογνώμονες ε, θα το συζητήσουμε, αλλά προσπαθήσουμε να πιέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Είμαι ευγνώμων, λέει ο πρόεδρο, γιατί τότε θα πρέπει να λάβουμε απόφαση όταν ε, θα ακούσουμε του επιρογνώμονες. Το είπα τέσσερις φορέ ήδη. Κύριε Καλιάκο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για όλα τα σχόλια που άκουσα. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντική η συζήτηση. Θα ήθελα να ε, πω ορισμένα πράγματα και βεβαίως ε, εγώ στην ε, Επιτροπή θα μεταφέρω όλα όσα άκουσα. Καταρχάς θα ήθελα να υπενθυμίσω τις απαρχές του κανόνα. Ο κανόνας εγκρίθηκε μετά από μια σοβαρή τρομοκρατική απειλή, η οποία είχε ως αποτέλεσμα ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο Ε, τώρα γνωρίζουμε τι ακριβώς έγινε. Ε, υπήρχε μια συνωμοσία που θα επηρέαζε 7 αεροσκάφη με εκρηκτικά υγρά. Τέλος πάντων τώρα το γνωρίζουμε, τότε δεν το ξέραμε. Ήταν λοιπόν μία ε, απειλή ε, κατά της ασφαλείας, η οποία εξακολουθεί να υφίσταται όμως και στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου που έχουν εγκρίνει τον ίδιο κανόνα. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο, είναι στόχος μας να προσπαθήσουμε να τον αλλάξουμε το συντομότερο δυνατόν. Να μειώσουμε όσο το δυνατόν ε, την δυσκολία για τους επιβάτες, το, την ε, ύπαρξη ενός καλύτερου συστήματος, ε, γιατί κανένας δεν το συμπαθεί αυτό το σύστημα, αλλά είναι ένας κανόνας που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως είπα υπάρχουν και σε άλλα μέρη του κόσμου αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η απειλή. Τρίτον, γεγονός είναι ότι οι πληροφορίες που λάβαμε είναι ότι μέχρι το 2010 θα είχαμε την, ε, τον τεχνολογικό εξοπλισμό στη διάθεσή μας και πρέπει να πω, πρέπει να το αναγνωρίσω ότι οι πληροφορίες που έχουμε και από τα κρατημέλη και από τους κατασκευαστές, από όλους, ότι υπάρχει περιπτώσει η τεχνολογία αυτή δεν είναι διαθέσιμη ακόμη ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε στις Ηνωμένε Πολιτείες, πουθενά. Άρα αυτό ήταν ένα σφάλμα το οποίο κάναμε και εμείς, αλλά και όλοι, όλες οι υπόλοιπε χώρες ε, που έχουν ε, τον συγκεκριμένο κανόνα ενισχύει. Συγγνώμη, Εν πάση περιπτώσει, και εμεί θα θέλαμε το 2010 να τα είχαμε έτοιμα όλα και να τελειώσει αυτό το πρόβλημα. Τώρα είναι έτοιμε οι Ηνωμένε Πολιτείε. Οι Ηνωμένε Πολιτείε θα κάνουν δοκιμέ για του επόμενου 18 μήνε. Κανένα δεν είναι έτοιμο ακόμη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, τι γίνεται με την τεχνολογία. Νομίζω ότι ο, Σίμσον, ο Σίμψον το εξήγησε πολύ καλά. Υπάρχουν τέσσερα είδη τεχνολογίας, ε, τύπος α, ανοίγει κανείς ε, το μπουκάλι, ελέγχει αν είναι κρυκτικό, αλλά πρέπει να το κάνει για το κάθε μπουκάλι. Δεύτερον, δεν ανοίγει το μπουκάλι, αλλά το βάζει μέσα σε, μια, σε ένα μηχάνημα. Ο, το type, ο τύπος ε, είναι αυτός που έχουμε τώρα, που μπορεί να βαθμιστεί και αυτό, είναι, αυτό το μηχάνημα έχει τα πιο υποσχόμενα αποτελέσματα και το ο τύπος Δέλτα είναι ε, ότι απλώς τα ελέγχουμε χωρίς να τα βγάλουμε από τις αποσκευές αυτό. Έχουμε πολύ χρόνο ακόμη μέχρι να είναι διαθέσιμο. Ε, και δεν θα το έχουμε σύντομα, εν πάση περιπτώσει. Τι προτείνουμε τώρα, και είναι κάτι που πρέπει βέβαια να το συζητήσουν οι εμπειρογνώμονε. Σωστό είναι αυτό, οι εμπειρογνώμονε. Ποια είναι η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτον, να βρούμε μια λύση για του επιβάτε σε τράνσιτ. Να μην γίνεται κατάσχεση. Να τελειώσει αυτό, να σταματήσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνουμε αυτό. Ε, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή οι τράνζιτ επιβάτε από τρίτε χώρε. ε, ε δεν, δεν μπορούν να κρατήσουν τα υγρά αυτά που έχουν στην κατοχή τους, κατάσχονται. Γιατί εκτός αν υπάρχει βέβαια κάποια διεθνή συμφωνία, αλλά... Ε, εν πάση περιπτώσει, κάποια αεροδρόμια μπορούν να πούν έρχεται από την Κροατία, έρχεται από τη Σιγκαπούρη και υπάρχουν κάποιε διαφορέ. Εμεί λοιπόν προτείνουμε οι επιβάτε transit να μην υπόκεινται σε αυτή τη διαδικασία κατάσχεση και προσπαθούμε ε, να, ζητήσουμε να συμφωνήσουμε με τα κράτη-μέλη που μας ζητούν να διορθώσουμε κάπως την κατάσταση. Δεύτερον, προτείνουμε μέχρι το 2012 να βρεθεί μια λύση για τα πιο σημαντικά αεροδρόμια. Νομίζω ότι μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Θα το συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη. Τώρα, χρειάζεται. Εντάξει, τα μικρότερα δρόμια μπορούν να φτάσουμε μέχρι το 2014 αν χρειάζονται, δύο ακόμα χρόνια. Μπορούν να γίνουν ε, νωρίτερα όλα αυτά δεν ξέρω. Αν μπορέσουμε ευχαρίστως, αλλά πρέπει να γίνει υπεύθυνα και με έλεγχο. Δεν μπορούμε απλώς ε, να μεταφέρουμε τις ημερομηνίες ε, αν ε, απλώς για να λέμε ότι το κάναμε νωρίτερα. Θα πω βέβαια στους εμπειρογνώμονες ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια συγκεκριμένη ημερομηνία την οποία να μπορούμε να τηρήσουμε. Επίσης, αυτές είναι τελικές. Τελικές ημερομηνίες. Είναι το αργότερο βέβαια θα υπάρχει ένα κίνητρο Οπότε, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να, ε, μας να, ενημε, να ενημερώσει ότι κάποια αεροδρόμια μπορεί να περάσουν στο επόμενο σύστημα, κάτι το οποίο βέβαια ως κίνητρο μπορεί να οθήσει κάποιους να μπορέσουν να εξεύρουν μια λύση νωρίτερα. Θα υπάρχει μια δυνατότητα αναθεώρηση, αν υπάρχει ένα διεθνές σύστημα για παράδειγμα, αν ε, το κάνουν πρώτε οι Ηνωμένε Πολιτείε, εμείς δεν θα πούμε όχι θα καθυστερήσουμε την κατάσταση. Αν υπάρξει ένα διεθνές σύστημα το οποίο ε, μπορεί να εφαρμοστεί. Εμείς είμαστε σε στενή επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το συζητούμε μαζί τους, είμαστε και πρωτοστάτες ε, στην, στον τομέα αυτό. Πιέζουμε και άλλες χώρες που είναι πιο επιφυλακτικές, που λένε ότι εν πάση περιπτώσει έχουμε ένα σύστημα, να το διατηρήσουμε, το έχουν συνηθίσει οι επιβάτες. Εμείς δεν θεωρούμε ότι αυτή είναι η λύση. Όχι, πρέπει να ζητήσουμε, να αναζητήσουμε μια λύση που να βασίζεται στην προηγμένη τεχνολογία του στο μότερο δυνατόν. Τώρα, Υπάρχει σημαντική πρόοδος ε, όσον αφορά το, την τεχνολογία. Οι κατασκευαστές ε, κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά πρέπει να υπάρχει σαφήνεια. Αυτός ο κανόνας για πάντα θα ισχύει. Ε, πρέπει να θέσουμε μία ημερομηνία κάποια στιγμή, γιατί αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να είμαστε πιο σαφείς, να γνωρίζουμε πότε θα γίνει η πώληση ε, της ε, εν λόγω τεχνολογίας και πότε μπορούν τα κράτη-μέλη να τη χρησιμοποιήσουν, να τη θέσουν σε εφαρμογή. Αυτή είναι η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Και θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας κάτι πολύ σημαντικό που το είπε και ο Πρόεδρος. Εμείς Κοιτάξτε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει το δικαίωμα γνωμοδότησης για το τελικό ε, σύστημα που θα εφαρμοστεί, γιατί είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί με του εμπειρογνώμονε ασφαλεία. 18 Νοεμβρίου θα γίνει μια συζήτηση στην διαδικασία επιτροπολογία, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιτροπολογίας. Μετά θα, γίνει μια, θα υπάρξει μια προθεσμία τριών μηνών που... Ε, εντός της οποίας το Κοινοβούλιο μπορεί να πει αν συμφωνεί, αν είναι αυτή η κατάλληλη διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας, γιατί εμείς δεν θέλουμε να γίνει απόρρεψη, θέλουμε να λάβουμε υπόψη τα σχόλια τα οποία άκουσα και να έχουμε όσο το δυνατόν την καλύτερη ε, τεχνολογική λύση. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώς θα, μειωθεί, πώς θα μειωθούν οι ουρές, πώς θα είναι με καλύτερη η κίνηση, ε, να επισπεύσουμε κάπως τη διαδικασία. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένας κανόνας, ένα σύστημα. Αν το σύστημα δεν ε, είναι διαθέσιμο και αν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, θα πρέπει, θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και γι' αυτό ακριβώς ε, ο Επίτροπος Ταϊάννη επέμεινε πριν συνεδριάσει η Επιτροπή των Εμπειρογνωμών, να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων ε, μεταξύ ημών και ημών, κάτι το οποίο εμείς πραγματικά εκτιμούμε όλους ιδιαίτερως, γιατί μας δώσατε πάρα πολλά στοιχεία που αξίζουν τον κόπο να τα λάβουμε υπόψη. Εγώ θα τα ε, μεταφέρω στους εμπειρογνώμονες. Είναι πάρα πολύ σημαντική μια εξισορροπημένη λύση για τη βελτίωση της παρούσας κατάστασης, όπως είπαν και οι περισσότεροι ε, συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η παρουσίαση σημειώματος ενημερωτικού για τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης επί του τομέα μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Κυρία Μαρκάλιο και τον κύριο Βάντεν Βόρντ έχουμε. Foster. Κυρία Φώστερ. Um, Συγγνώμη που διακόπτω. Δεν είδαμε τον ημερωτικό σημείωμα. Προσπαθήσαμε να το βρούμε. Και μας είπαν ότι δεν είναι διαθέσιμο. Και δεν είναι διαθέσιμο μέχρι τη συνεδρίαση. Εγώ δεν είδα τίποτα σαν μέλος της Επιτροπής αυτής. Θα, μοιραστεί τώρα αυτή η μελέτη, έρχεται. Δεν ξέρω πότε ετοιμάστηκε. Για να γίνει μια παρουσίαση της έκθεσής τους. point of Διαδικαστικό, προσπαθούν να ετοιμάσουν κάτι. Θέλω να κάνω μια παρουσίαση στην Επιτροπή αυτή. Θέλω να συζητήσω με ένα ενημερωτικό σημείωμα να εκφράσουν απόψει. Όταν πηγαίνει κανείς στην Επιτροπή, ίσως κάποια μέλη θέλουν να σχολιάσουν σχετικά με τα υποθέντα και ε, δεν έχει νόημα να μοιράζεται το ενημερωτικό σημείωμα ενώ η συζήτηση ξεκινά. Ζητήσαμε να κάνει κάτι η γραμματεία και εσείς σαν πρόεδρος Επιτροπής παρακαλώ να υπενθυμίσετε σε όσου θέλουν να συζητηθεί κάτι εδώ να δίνει τουλάχιστον την προηγούμενη το πρωί αν γίνεται η συζήτηση το απόγευμα, να δίνετε το έγγραφο. Fruitful discussion. Thank you, Chairman. Το λαμβάνω υπόψη, λέει ο Πρόεδρος. Θα το διαβιβάσω στην Γραμματεία. Ούτως στο μέλλον, οσδήποτε κάνει παρουσίαση στην Επιτροπή, να δίνει την παρουσίαση αυτή στα μέλη εκ των προτέρων. Και όχι ένα λεπτό πριν ξεκινήσουμε, δεν είναι ο προηγουμένος ένα λεπτό μόνο. Ετέφη. Ξεκινάει η παρουσίαση. Maybe better go on the, the two on the end, yeah. 15 λεπτά ας πούμε για την παρουσίαση θα χρειαστούμε. Και μετά θα υποβληθούν ερωτήσεις, θα ακουστούν σχόλια και ελπίζω τα μέλη να έχουν το χρόνο να διαβάσουν λίγο το έγραφο αυτό. We're ready when you are. Okay need to press the button to put the microphone on. Oké, okay, hartelijk uh, dank voorzitter voor uh, de kans om onze briefingnota hier te komen voorstellen. Ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσουμε το ενημερωτικό μας σημείωμα. Θα το κάνουμε σύντομα και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε και σε ερωτήσεις που τυχόν να έχετε. Τώρα, να σας πω τι ακριβώς, ε, σε τι ακριβώς έγκυται. Έχει πέντε τμήματα η παρουσίαση μας. Μισό λεπτό διακόπτει ο πρόεδρος. Αν δεν θέλετε να δείτε την παρουσίαση και θέλετε να συζητήσετε, παρακαλώ να βγείτε από την αίθουσα. Δεν γίνεται να έχουμε τρει-τέσσερι παράλληλε συναντήσει. Αν θέλετε να μιλήσετε, να βγείτε έξω από την αίθουσα. Συγγνώμη που σα διακόψα, λέει ο πρόεδρο. Ευχαριστώ. Βλέπετε λοιπόν ε, το περιεχόμενο της έκθεσης, εισαγωγή, να πω ορισμένα πράγματα για τη δομή της, ε, των εναέριων μεταφορών. Ε, δεν πρέπει να το θεωρείτε ένα ενιαίο προϊόν. Μετά θα δούμε τάσεις από το παρελθόν μέχρι πολύ προσφάτως και μετά θα προσπαθήσω να σας πω ορισμένα πράγματα για τον αντίκτυπο της κρίσης και να σας πω Ποιε ακριβώ ήταν οι συνέπειες. Θα κάνουμε στη συνέχεια κάποιε προτάσει. Αν δει κανεί τις συνέπειες της κρίσης, τα ακούσαμε λίγο και στην ε, περασμένη συζήτηση που είχαμε κάνει. Πρώτον, Υπάρχει ε, μια σοβαρή μείωση στις ε, εναέριες μεταφορές. Πολλές ε, αεροπορικές εταιρείες το είχαν προβλέψει αυτό και είχαν μειώσει τον αριθμό πτήσεων που προσέφεραν. Από 15% έως 25% ήταν η μείωση αυτή. Αλλά δεν ήταν τόσο πολύ σημαντική η μείωση αυτή. δηλαδή, ροές μεταφορών δεν έχουν αλλάξει τόσο πολύ. Γιατί μερικά δρομολόγια συγχωνεύτηκαν, για παράδειγμα. Επίσης βλέπετε τον αντίκτυπο της κρίσης ε, στα κέρδη. Σοβαρή μείωση. Έχουν μειωθεί πολύ λοιπόν τα κέρδη των ε, εταιριών και επίσης ε, έχουν αλλάξει και οι στρατηγικές μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση στο μέλλον λόγω της κατάστασης αυτής. Μάλιστα. Απλώς για να σας πω ποιος συμμετέχει στην όλη διαδικασία, πώς μπορούμε να συσχετίσουμε τα πράγματα. Γνωρίζετε ότι η κρίση αυτή τη στιγμή είχε ως αποτέλεσμα μείωση της επιβατικής κίνησης κατά 15 έως 25% και αυτά είναι στοιχεία που μας δίνει ο ίδιος ο κλάδος των μεταφορών. Όλα αυτά είναι ποικιλίε ουσιαστικά στοιχείων που είναι αποφασιστικές για να μας εξηγήσουν ποια είναι η εξέλιξη στον τομέα των μεταφορών. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη σχέση μεταξύ της βιομηχανικής παραγωγής και του, των ε, λιανικών πωλήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτές λοιπόν ε, οι καμπύλες έχουν αυτές οι διακυμάνσεις έχουν επηρεάσει ιδιαίτερα την ανάπτυξη των αεροπορικών εμπορευματικών μεταφορών. Ενώ στο παρελθόν δηλαδή οι αεροπορικές μεταφορές ακολουθούσαν τους οικονομικούς κύκλους, δηλαδή την εξέλιξη του ΑΕΠ, βλέπουμε ότι πια δεν υπάρχει μια τέτοια σύνδεση, αλλά υπάρχει περισσότερο μια σύνδεση με, τις, ε, με τον όγκο των λιανικών πωλήσεων και με την συνολική βιομηχανική παραγωγή. Next slide, please. Σε αυτή τη διαφάνεια, αυτό το οποίο μπορούμε να δούμε είναι το ποσοστό πληρότητος για τις πτήσεις των εταιριών ΣΥΑΤΑ και ποιες είναι οι εξελίξεις 2009 έναντι του 2008 για διαφορετικές περιοχές του κόσμου, γεωγραφικές περιοχές φυσικά, και βλέπουμε πώς αυξήθηκαν τα έσοδα ανά χιλιόμετρο για τις αεροπορικές εταιρείες και βλέπουμε και τον, ε, τον παράγοντα πληρότητος για τις ε, εταιρείες αυτές. Βλέπουμε επίσης ποια είναι η αύξηση του βάρους που μεταφέρεται ανά χιλιόμετρο και επίσης και του, της προσφοράς χωρητικότητας από τις εταιρείες. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μία απώλεια από το 2008 ως το 2009 της τάξης των 7,6% κατά μέσον όρο σε επίπεδο παγκόσμιο, δηλαδή σε έσοδα ανά επιβάτη σε παγκόσμιο επίπεδο και περίπου 3,9% μείωση σε συνολικά έσοδα. Ο παράγων πληρότητος εξακολουθεί να είναι παρά αυτή τη μείωση των εσόδων σε ένα καλό επίπεδο στα 72,6%. Πρέπει εδώ να υπογραμμίσουμε ότι οι περιοχές του κόσμου όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη ανάπτυξη είναι εκεί που υπάρχουν οι φέτες ηλικία που ταξιδεύουν περισσότερο, δηλαδή οι ηλικίε που ταξιδεύουν περισσότερο, εκεί υπάρχει μεγαλύτερη μείωση των εσόδων. Αλλά υπάρχει και μια μεγάλη, μεγάλη διαφορά μεταξύ της ε, εξέλιξη στις αγορές ε, επιβατών, στην επιβατική αγορά και στην αγορά των εμπορευμάτων. Έχουμε περίπου μείον 20% σε ό,τι αφορά τα, τους τόνους χιλιόμετρα, ενώ για τους επιβάτες είναι μονάχα 7,6 μείωση. Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο αυτών αγορών, που όπως είπαμε προηγουμένως είναι οι αγορές που συναγωνίζονται για τα ίδια ουσιαστικά αεροσκάφη. Βλέπουμε λοιπόν την σημασία του μικτού χαρακτήρα των αεροπορικών μεταφορών και που βασίζονται κυρίως στις, ε, ε, σε δύο διαφορετικές αγορές με μικρή μοναχα επικάλυψη των δύο. Η επόμενη διαφάνεια. Εδώ βλέπουμε την ε, τροποποίηση του ΑΕΠ από το 1990 έως το 2008 για διάφορες περιοχές του κόσμου, Ιαπωνία, Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέπετε ότι υπάρχει μία παρακολούθηση κατά κάποιο τρόπο από την ε, αεροπορική βιομηχανία του ΑΕΠ των σημαντικών αυτών περιοχών. Δηλαδή η αύξηση των αεροπορικών μεταφορών αντιστοιχεί στην ε, αύξηση του ΑΕΠ αντιστοιχούσε, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή ανατρέπεται όπως σας έδειξα στις προηγούμενες διαφάνειες. Η ανάλυση τώρα της κρίσης. Έχουμε ένα σύνολο φαινομένων τα οποία παρατηρήθηκαν, μια σειρά από οι οποίες αναδύονται. Οι περισσότερες από αυτές τις τάσεις δεν έχουν ξεκινήσει με την οικονομική κρίση και θα πρέπει να δούμε τώρα <clears throat> ποια είναι τα στοιχεία τα οποία ενισχύθηκαν ιδιαίτερα λόγω της κρίσης. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να δούμε ποια είναι τα φαινόμενα τα οποία έχουν καθορίσει την εξέλιξη ε, των αεροπορικών μεταφορών. Οι συγχωνεύσεις, η παγιοποίηση και η κάλυψη των μικρών αγορών, δηλαδή η στατηγική των αεροπορικών εταιριών και ο τρόπος με τον οποίο προσπαθήσανε να κατακτήσουν περισσότερες αγορές στη σειρά των διαφόρων κρίσεων που είχαν αποτελέσματα στους πόρους του τομέα αυτού. Υπάρχει το θέμα της ιδιωτικοποίησης και το τέλος των εθνικών αεροπορικών εταιριών. Είναι ένας από τους κύριους παράγοντες, μια από τι μεγαλύτερες αλλαγές που έχει λάβει η χώρα τα τελευταία χρόνια στην αεροπορική βιομηχανία. Και εδώ υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία σε ό,τι αφορά την κρατική συμμετοχή στις επιχειρήσεις, τι αεροπορικέ. Επίσης, η σημασία των διασταυρούμενων συγχωνεύσεων ή εξαγορών μεταξύ ε, εταιριών διαφόρων χωρών και οι συμμαχίες μεταξύ εταιριών που βρίσκονται σε διάφορες χώρες τίθεται και σε αμφισβήτηση το μοντέλο το οποίο είναι γνωστό ως μοντέλο Southwest, δηλαδή το μοντέλο των φτηνών εταιριών, εταιριών χαμηλού κόστους, γιατί και αυτό το υπόδειγμα αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται από την οικονομική κρίση. Έχουμε φυσικά μεγαλύτερο αριθμό πτωχεύσεων, λόγω της ίδιας της, της δυναμικής της ε, κρίσης έχει επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία των ε, πτωχεύσεων αεροπορικών εταιριών και επηρεάζει την είσοδο και την έξοδο από την αεροπορική αγορά. Παραμένει πάρα πολύ δυναμικός ο τομέας αυτός. Ενώ αυξήθηκε ο αριθμός των πτωχεύσεων, αυξήθηκε ο αριθμός των νέων εταιριών και υπάρχει μια μεγαλύτερη επιθετικότητα στον εμπορικό τομέα με πιο εφάνταστες τεχνικές marketing. Φυσικά αλλάζει και η επιρροή των κυβερνήσεων που έχουν μεγαλύτερη επιρροή και μικρότερη μάλλον επιρροή και μικρότερη παρέμβαση στην αγορά εφόσον δεν υπάρχουν πια οι εθνικές εταιρείε και έχουμε μια τεράστια διακύμανση στην αγορά, μια μεγάλη αστάθεια και διακύμανση στην αγορά των εμπορευμάτων, της μεταφοράς εμπορευμάτων που υπάρχει και η τάση να μεταφέρονται σε ειδικευμένε εταιρείε οι οποίες δεν συμπίπτουν πάντα με τις εταιρείε επιβατηγών μεταφορών. Υπάρχει όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή ξένου κεφαλαίου και φυσικά με όλη αυτή τη δυναμική, με όλη αυτή τη διαδικασία πτωχεύσεων και το άνοιγμα <clears throat> νέων ε, τομέων και νέων εταιριών, βλέπουμε <clears throat> ότι μειώνεται και η απασχόληση στον τομέα αυτό και προκύπτουν και κάποιες εταιρείε οι οποίες είναι μεσάζοντες για την παροχή ειδικευμένων θέσεων εργασίας. Επόμενη διαφάνεια. Βλέπουμε εδώ πέρα την ε, απώλεια θέσεων απασχόλησης η οποία έγινε μέσα στον τελευταίο χρόνο. Η SAS ε, απέλησε περίπου το 1 τρίτο των εργαζομένων, τους 8.600 από 23.000 και τον Αύγουστο του έτους αυτού ακόμα 1.000 με 1.500 θέσει εργασία απολέτησε. Η Virgin Atlantic τον Φεβρουάριο ε, περιέκοψε 600 θέσει από 9.000, η Ryanair 200 <clears throat> το Φεβρουάριο, η Air France 3.000 τον Απρίλιο από 100.000 που μπορεί να φτάσουν και 100.000 τα επόμενα χρόνια. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι μόνο οι παλιές εθνικές εταιρείες οι οποίες περικόπτουν θέσει εργασία, αλλά πολλέ φορέ και μερικέ από τι νέε εταιρείε, ακόμα και οι εταιρείε χαμηλού κόστου, όπω η διαβόητη Ryan και Air. Επόμενη διαφάνεια. Ευχαριστώ. Έχουμε τρεις διαφάνειες εδώ που τις ετοιμάσαμε για να σας δείξουμε κάποια σημαντικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να ελεγχθούν. Αριστερά βλέπουμε το θέμα στην αριστερή στήλη μετά έχουμε ενδεχόμενες συνέπειες και μετά βλέπουμε τις συνέπειες της κρίσης. Εδώ έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες από ό,τι στο ενημερωτικό ε, σημείωμα. Έχουμε εδώ τις συμμαχίες ε, και τους διάφορους βασικούς πρωταγωνιστές, αν θέλετε, στον τομέα. Συγκέντρωση που δημιουργεί κίνδυνο ότι μακροπρόθεσμα μπορούμε να έχουμε κάποια δεσπόζουσα θέση στην αγορά και κατάχρηση αυτής της δεσπόζουσας θέσης. Όχι γενικά, αλλά για κάποια δρομολόγια. Ποιες είναι οι συνέπειες της κρίσης. Λόγω των εξελίξεων και την ανάγκη ανακεφαλαιοποίησεως κάποιων αεροπορικών εταιριών και πιο συγκεκριμένα το κεφάλαιο των μεγαλύτερων ομίλων, βλέπουμε ότι η ενοποίηση προχωρά με ταχύτερους ρυθμούς Ταυτόχρονα, σαν αποτέλεσμα της κρίσης, είναι πολύ δύσκολο να φτιάξεις μια αεροπορική εταιρεία για κάποιο συγκεκριμένο δρομολόγιο. Χρειάζεσαι, κρίσιμη μάζα. Το τελευταίο τρίμηνο, ο αριθμός των αεροπορικών εταιριών, πολλές εταιρείε που άνοιξαν ξεκίνησαν. Υπήρχε διασύνδεση Αμβέρσας Φραγκφούρτης, κράτησε δύο-τρεις μήνε και έκλεισε. Μετά, δεύτερο σημείο, ιδιωτικοποίηση και το μερίδιο το κρατικό στον τομέα, το ποσοστό. Παρόμοιες τάσεις διαπιστώνουμε. Ε, η, τρίτη φορής, αν θέλετε, για τις υπηρεσίες που παρέχουν, υπεργολαβεί όσον αφορά τις υπηρεσίες εδάφους. Και εκεί βλέπετε μια μετακίνηση προς ενοποίηση και συγκέντρωση. Επίσης, είδαμε τι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και βλέπουμε ότι υπάρχουν μόνο 6-7 ανταγωνιστές στην ευρωπαϊκή αγορά. Αν δείτε εξαγορές και συγχωνεύσεις δεσυνοριακά, αυξάνεται η τάση Lufthansa παραδείγματος χάρη, η οποία Lufthansa αγοράζει μετοχές σε μικρότερες εταιρείες και αυτό οδηγεί σε ενοποίηση. Όλα αυτά επιταχύνονται λόγω της κρίσης. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα πέρα από τη Λουφτχάντσα. Και η στρατηγική της Λουφτχάντσα δεν είναι παντού ίδια. Η παραδείγματη. Έχουμε την Swiss στη Ζηρίχη που προσπαστεί να εστιαστεί προσπαθεί να εισαχθεί η Lufthansa σε τρει εταιρείε ελβετικές μεταξύ των οποίων ε, ε, η Swiss, αλλά δεν κάνουν το ίδιο με την BMI και με άλλε εταιρείε. Μετά οι εταιρείε χαμηλού κόστου. Εκεί οι μικρότερε εταιρείε εξαφανίζονται και εκεί βλέπουμε συγκέντρωση περιορισμένο αριθμό μεγάλων εταιριών, Ryanair είναι ένα παράδειγμα, και αυτή η τάση συνεχίζεται και επιταχύνεται. Και αυτό που συνέβη πρόσφατα, και είναι σημαντική τάση αυτή, είναι αυτό που ανέφερε η Ροζάρια, ότι τα όρια μεταξύ της εταιρείας χαμηλού κόστους και των άλλων αεροπορικών εταιριών ε, γίνεται όλο και πιο θολή. Η Ryanair, Φερρυπίν. Και ποια τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος χαμηλού κόστους. Mm. Αλλάζει η Ryanair ε, έχει όλο και περισσότερε πτήσει μεγάλης απόσταση, α πούμε Βρυξέλλες, Τενερίφη και προσπαθεί να συναγωνιστεί με τις εταιρείε charter και να διεκδικήσει νέες αγορε. Χρεοκοπίες. Κατανοητό ότι θα συνεχιστεί η τάση και για τους επόμενους μήνες σαν αποτέλεσμα υποτονικής κεφαλοποίησεως κάποιων μεγάλων εταιριών υπάρχουν συνέπειες όπως ενοποίηση, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος της δημιουργίας δεσπόζουσας θέσης στην αγορά και κατάχρησης αυτής. Τέλος τη διαφάνεια, τελευταία γραμμή είναι οι νέες εταιρείε στην αγορά. Πιθανότατα στο μέλλον θα είναι πιο εύκολο για μια νέα εταιρεία να χρησιμοποιήσει στρατηγικές όπως πολύ χαμηλές τιμές για να ισχυροποιηθεί και να η μάλλον παλιά εταιρεία να ρίξει πολύ τις τιμές για να προσπαθήσει να κρατήσει εκτός τις νέες εταιρείε. Και τώρα σε αυτή τη διαφάνεια δείχνουμε μερικές από τις πιο σημαντικές εξελίξεις στον τομέα αυτό της ε, αεροπορικής βιομηχανίας, η εισαγωγή των συστημάτων εμπορίας εκπομπών και με τον τρόπο αυτό πέναμε σε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έχει να κάνει με την βιωσιμότητα των μεταφορών. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για την κοινωνία μας, γιατί ξέρουμε ότι και οι αεροπορικές εταιρείες είναι από τους κύριους που ρηπαίνουν και επομένως φύγουν την βιωσιμότητα του πλανήτη μας. Η οικονομική κρίση θα ενισχύσει αυτή τη διαδικασία γιατί από τη μία πλευρά επιταχύνει τη διαδικασία της εφαρμογής της αγοράς εκπομπών αλλά έχει σαν αποτέλεσμα αυτή η ίδια η εφαρμογή αυτού του συστήματος να έχει πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο στο, στη διάρθρωση κόστου των εταιριών. Επομένως θα είναι όλο και πιο μεγάλος ο αντίκτυπος αυτός και ο οποίος θα έχει έτσι κάποια αποτελέσματα, τουλάχιστον μπορούμε να προσδοκούμε να έχει αποτελέσματα στην τεχνολογική ε, εξέλιξη. Επομένως, οι στρατηγικές που θα ακολουθήσουν οι εταιρείε αυτές θα επηρεαστούν από την συνεργειακή δράση της εισαγωγής του εξωτερικού κόστους μέσα στα πλαίσια της κρίσης. Η αγορά των εμπορευμάτων, της μεταφοράς εμπορευμάτων είναι μια αγορά που διέρχεται μεγάλες αλλαγές και ένα από τα αποτελέσματα αυτής της κρίσης είναι το γεγονός ότι έχει κατανοήσει η αεροπορική βιομηχανία ότι ακριβώς λόγω των αποτελεσμάτων της οικονομικής κρίσης είναι απαραίτητο να υπάρξει μια εταιρική σχέση των ε, εμπορευματικών μεταφορών με άλλους τρόπους μεταφοράς εμπορευμάτων. Αυτό έχει επηρεάσει λοιπόν τις αγορές και αυτό ίσως θα τροποποιήσει περισσότερο την αγορά εμπορευματικών αεροπορικών μεταφορών, ότι θα υπάρχει λοιπόν μεγαλύτερη και εταιρικότερη σχέση με τους άλλους τρόπους μεταφορών και θα είναι μονάχα ένας μεταξύ πολλών τρόπων μεταφορών η αεροπορική οδός. Είναι σαφές ότι αυτό σημαίνει μια μεγαλύτερη κατανομή ε, σε σχέση με τις εταιρείε που είναι καθαρά εμπορευματικές και τις εταιρείε που είναι επιβατικές και μεταφέρουν και ε, εμπορεύματα, θα προσπαθήσουν οι εταιρείε λοιπόν να αποσπάσουν το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος για να μπορέσουν με τον τρόπο αυτό μέσω των εμπορευματικών μεταφορών να χρηματοδοτήσουν και τις επιβατικές μεταφορές. Χάρη λοιπόν σε εμπορευματικές μεταφορές μπορούν να χρηματοδοτούν τον τομέα επιβατών και να είναι πιο επιθετικοί στον τομέα αυτών των επιβατών. Όλα αυτά λοιπόν είναι μια επιτάχυνση τη διαδικασία αυτή λόγω τη κρίσεω. Υπάρχει μεγαλύτερη φαντασία, μεγαλύτερη επιθετικότητα και οι οικονομικοί φορεί προσπαθούν να προχωρήσουν και προ μια κατεύθυνση μεγαλύτερη οικονομική συγκέντρωση, μεγαλύτερη κτίση μεριδίου τη αγορά, ώστε να μπορέσουν να σταθεροποιήσουν την πηγή εσόδου του. Λόγω αυτή τη κρίση. αυτή η στρατηγική θα του οδηγήσει έξω από τα σύνορα τη αεροπορική. Ε, του αεροπορικού τομέα και επομένως θα προχωρήσουν και σε συγκέντρωση αγοράς σε ευρύτερο επίπεδο. Υπάρχει μια ένταση και εντατικοποίηση ξένου κεφαλαίου σε αυτές τις επιχειρήσεις και επομένως υπάρχει ο κίνδυνος να υπάρξει υπερσυγκέντρωση κεφαλαίου σε ένα περιορισμένο <clears throat> αριθμό ισχυρών ομήλων, οι οποίοι μπορούν έτσι να ελέγξουν ένα σύνολο από κρίσιμα δίκτυα μεταφορών σε σχέση με τις εναέρειες μεταφορές. Μπορεί λοιπόν να καταλήξουμε σε μια κατάσταση δεσπόζουσας θέσης που στη συνέχεια θα οδηγήσουν σε κυριαρχικού χαρακτήρα στρατηγικές. Αυτό έχει συμβεί σε άλλους τρόπους μεταφοράς και επομένως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα αποτελέσματα αυτής της παρουσίας του κεφαλαίου που είναι πιο έντονη από ό,τι σε άλλες στρατηγικές αγοράς. Επομένως θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε άλλα εργαλεία για την παρακολούθηση των αγορών της, ε, του αεροπορικού τομέα. Καταλήγουμε λοιπόν στο πρώτο next slide, στο πρώτο συμπέρασμά μας. Πράγματι, η αλλαγή η οποία έχει γίνει στον τομέα της αεροπορικής βιομηχανίας και γενικά σε όλο τον τομέα των ενέργειων μεταφορών, έχει σαν αποτέλεσμα να τροποποιούνται οι αγορές και να τροποποιούνται και οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι φορείς με έναν τρόπο υπερβολικά και έντονα δυναμικό. Κάτι το οποίο βλέπουμε λοιπόν ότι πρέπει να ασκηθεί η ρυθμιστική λειτουργία πολλές φορές με ένα τρόπο κατασταλτικό με την επιβολή κυρώσεων στους κακούς, αλλά συγχρόνως δεν δίνει τη δυνατότητα στο ρυθμιστικό, στις ρυθμιστικές αρχές να ακολουθούν μια στρατηγική προσέγγιση για να μπορέσουν να δώσουν κίνητρα για μια σωστή συμπεριφορά μεταξύ των καλών φορέων. Επομένως, αυτή τη στιγμή αντιδρά η ρύθμιση και δεν είναι ε, αυτοί οι οποίοι ανοίγει δρόμους για το μέλλον. Είναι σημαντικό λοιπόν να λάβουμε υπόψη την ανάγκη μιας παρακολούθησης η οποία θα πρέπει να γίνεται με ένα διαφορετικό τρόπο και όχι μονάχα με κατασταλτικό και τιμωρητικό χαρακτήρα. Εξάλλου, δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε οι διάφορες αγορές και υποαγορές και υποϊποαγορές εναερίων μεταφορών να παγιοποιηθούν και να συγκεντρωθούν σε στα χέρια μονάχα μερικών φορέων. Αυτή είναι και η, Αυτή είναι και η λογική της αγοράς. Αλλά αυτή η διαδικασία είναι μια φυσική διεργασία που οφείλεται στο ένστικτο αυτοσυντήρησης των εταιριών. Αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Αυτό όμως το οποίο είναι απαραίτητο σε επίπεδο παρακολούθησης είναι να υπάρχει εγκαίρως η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτών των συγκεντρώσεων. Επομένως, εμείς συμβάλλουμε, συμβουλεύουμε τις ευρωπαϊκές αρχές να παρακολουθήσουν και να benchmarkάρουν τις αγορές τις, ε, των ε, αερίων μεταφορών επί τη βάση των στοιχείων και της έρευνας που μπορεί να προέλθει από την παρακολούθηση αυτού του τομέα και δίνοντας την μεγαλύτερη δυνατή έμφαση στην παρακολούθηση της οικονομικο-βιομηχανικής συμπεριφοράς όλων των φορέων στον τομέα αυτό προοπτική να υπάρξει μια με στρατηγικό όραμα ρύθμιση στην περιοχή αυτή, η οποία δεν θα έχει καταστατικό μοναχα χαρακτήρα, αλλά θα οδηγεί και σε νέους ορίζοντες. Έτσι μπορούμε να κλείσουμε την ε, παρουσίασή μας και εξ του εαυτού μου και του κ. Βαντερβού. Σας ευχαριστούμε και είμαστε στη διάθεσή σα απολύτω για τα ερωτήματα τα οποία θέλετε θέση. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Mr. Κύριε Ελκαντράουι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, δεν πρόλαβα προφανώς να διαβάσω τη μελέτη σας, θα το κάνω όμως. Εν τω μεταξύ όμως ήθελα να κάνω τρεις ερωτήσεις και σχόλια. Είναι αλήθεια ότι η κρίση είναι πολύ χειρότερη αυτή τη φορά από την προηγούμενη το 2001 όταν υπήρχε και τότε κρίση στις αερομεταφορές. Σε μία από τις διαφάνειές σας μας δείξατε ότι έχουμε φτάσει στο χειρότερο επίπεδο. Έχουμε φτάσει στα χειρότερα επίπεδα. Βλέπω επίσης από τα αριθμιστικά, αριθμητικά σας στοιχεία ότι η Μέση Ανατολή είναι εξαίρεση. Εκεί υπάρχει αύξηση της κίνησης μεταξύ 2008 και 2009. Αυτό είναι φυσιολογικό. Είναι φυσιολογική η ανάπτυξη της αγοράς. Ενδεχομένως λόγω της ε, τράνζιτ επιβατικής κίνησης συμβαίνει αυτό. Και κάτι ακόμη. Το γενικό σας συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει κίνδυνο συγκέντρωσης και ότι αυτό μπορεί να έχει κακές συνέπειες. Αλλά εγώ νόμιζα ότι υπήρχαν ε, κάποιες μεγάλες ε, συμμαχίες και υπήρχαν και κάποιες ε, αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους. Ούτως ή άλλως, οπότε πότε αρχίζουμε να μιλάμε για δεσπόζουσα θέση. Τέσσερις, πέντε, Πόσοι πρέπει να είναι, δηλαδή πότε πρέπει να αρχίσει να ε, αντιδρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πότε αρχίζει να υπάρχει πρόβλημα. Ίσως να μπορείτε να μου απαντήσετε σε κάποια από αυτά τα ερωτήματά μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δύο-τρεις ερωτήσεις να ακούσουμε μαζί και μετά θα δοθούν οι απαντήσεις. Βέβαια, λέει ο κ. Γκρός. Θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα το οποίο δεν είναι ερώτημα ευγενικό. Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να αντιμετωπίσει η κάθε επιτροπή μεταφορών. Πώς βλέπετε την ρύθμιση για τις χρονοθυρίδες στα σλότ μέσα σε αυτή την ανάλυση που μας παρουσιάσατε. Γιατί εμείς ίσως θα πρέπει να δούμε αν θέλουμε να επανεξετάσουμε αυτή την αρχή των χρονοθυρίδων. Πρέπει να το κάνουμε ή δεν πρέπει να το κάνουμε. Δεν ξέρω αν είναι η κατάλληλη στιγμή να σας ζητήσω μια συμβουλή για το θέμα αυτό. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση. Εγώ συνεχίζω αυτό που είπε ο συνάδελφος μου, ο κύριος Αλκ Χαντρουή. Είπατε ότι φυσικά θα πρέπει να αναπτύξουμε τα εργαλεία για να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν στρεβλώσεις στην αγορά ή ότι θα υπάρξει κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Ποια είναι τα εργαλεία για τα οποία αναφέρεστε. Αναφέρεστε στο μερίδιο αγοράς για ορισμένες περιοχές ή για ορισμένες, για ορισμένες διαδρομές. Ίσως αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει τις ευρωπαϊκές εταιρείες σε προβλήματα ή το βλέπετε με άλλο τρόπο. Το τελευταίο ερώτημα που θέλω να θέσω όταν βλέπω την εξέλιξη των εταιριών χαμηλού κόστους σε ό,τι αφορά και τα αεροσκάφη και για την, τους επιβάτες. Φαίνεται ότι έχουν αντέξει την κρίση καλύτερα από τις άλλες εταιρείες. Είναι αλήθεια αυτό ή όχι. Ανταποκρίνεται στην ανάλυση σας, κύριε Φώστα. Ευχαριστώ πολύ ε, ε, κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους προσκεκλημένους μας. Επιμένω ότι έπρεπε να μας είχατε δώσει νωρίτερα αυτό το λεπτομερές εγγραφό σας. Πώς είναι δυνατόν να μας ζητάτε να σχολιάσουμε τόσο λεπτομερή στατιστικά στοιχεία. Δεν είναι ο κατάλληλος τρόπος για να γίνονται τα πράγματα. Σελίδα 29. Έχετε ένα κατάλογο αεροπορικών εταιριών και τις περικοπές της θέσης απασχόλησης και η British Airlines, British Airways λέγεται και το λέω γιατί για αυτούς δούλευα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τέλος πάντων, ας δούμε Πώ έχουν τα πράγματα. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι παρόλε τι στατιστικέ, από ό,τι θυμάμαι, επειδή πάνω από 25 χρόνια, 30 χρόνια ε, ήμουν στον κλάδο αυτό, αν δούμε τα αεροδρόμια στην Ευρώπη, υπάρχουν περίπου 150 εκατομμύρια επιβάτες ε, που πέρασαν από τα αεροδρόμια κατά το 2008 ε, προφανώς υπάρχουν επαρκείς αεροπορικές εταιρείε οι οποίες ε, παρόλα αυτά έχουν πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση να αντιμετωπίσουν. Έχουν ε, αυξηθεί και οι τιμές των καυσίμων. Κάπως καλύτερη είναι η κατάσταση τώρα, αλλά γνωρίζαμε ότι είχαν φτάσει σε άκρα οι τιμέ ε, Και είναι υπερχρεωμένε όλες αυτές οι εταιρείε. Θέλω να πω το εξή. Ποιο είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών. Εμείς γιατί είμαστε εδώ, γιατί έχουμε αεροπορικές εταιρείες, αεροδρόμια στις εκλογικές μας περιφέρειες, έχουμε τους κατασκευαστές που πουλούν ε, τους, ε, τα αεροσκάφη στον, ε, στα, στις αεροπορικές εταιρείες και ολόκληρη αυτή η αλυσίδα καταραίει. Εγώ από ό,τι θυμάμαι είναι χειρότερη κατάσταση από την πετρελαϊκή κρίση του 1974. Μιλάμε για τη χειρότερη κρίση. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξη, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Προσπαθούμε να ανταγωνιστούμε ε, παγκοσμίω. Ε, συμφωνώ με ένα από τα συμπεράσματά σας ότι δεν είναι δυνατόν να εισαγάγουμε κυρώσεις ε, νομοθετικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα έχουν επιβλαβεί συνέπειες ε, στην ε, στο, στον κλάδο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει να είναι πραγματικά πολύ σοβαρό ε, σημείο, πολύ σοβαρή πτυχή για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το Συμβούλιο, όταν σκέφτονται τι θέλουν να κάνουν για τη σχετική νομοθεσία. Όσον αφορά λοιπόν την αλυσίδα διανομής ε, συζητήσαμε πάρα πολλές φορές τα πράγματα σε σχέση με το κόστος. Μιλήσαμε για τη μεταφορά υγρών σε σχέση με το κόστος, ε, την κρίση σε σχέση με το κόστος. Πάντοτε το κόστος είναι πάρα πολύ σημαντικό, είτε πρόκειται για κατασκευές, είτε πρόκειται για περικοπές θέσεων απασχόλησης. Πάντα καταλήγουμε στο κόστος. Πώς είναι λοιπόν, ε, πώς θα, πώς θα βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Αυτές είναι οι προκλήσεις. Εγώ δεν τα παίρνω όλα αυτά ελαφρά την καρδία είναι πραγματικά πάρα πολύ ανησυχητικά γιατί οι κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες ε, της ε, ε, το τομέα των αερομεταφορών είναι πάρα πολύ σημαντικός και είναι τεράστιες οι συνέπειες και έχουν πολύ μεγάλη σημασία στην ανταγωνιστικότητά μας, στην ανταγωνιστικότητό μας στον κόσμο όλο. Επα, επίσης, ε, οι μεταφορές εμπορευμάτων, μόνο, μόνο για τις, επιβατικές, ε, μεταφορές επιβατών μιλάμε, αλλά ξεχνάμε το πόσο μεγάλο ποσοστό ανήκει στις μεταφορές εμπορευμάτων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν που ήρθατε. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να τα εξετάσουμε λεπτομερέστερα τα πράγματα, οπότε Α τα έχουμε εκ των προτέρων για να έχουμε μια πιο επικοδομητική συζήτηση, γιατί είναι σοβαρή η συζήτηση αυτή. Και να δούμε ποια είναι τα βασικά σημεία για τα οποία η Επιτροπή Μεταφορών μπορεί πραγματικά να συμβάλλει. Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε να απαντήσετε σε αυτές τις ε, πρώτες τρεις ερωτήσεις και μετά να ακολουθήσουν άλλες τρεις ερωτήσεις. Ξεκινώ με το πρώτο ερώτημα, το οποίο συνδέεται με το πρόβλημα της κρίσης. Καταρχήν αυτή η κρίση δεν είναι χειρότερη από τις προηγούμενες. Αλλά προκύπτουν από αυτή χειρότερα αποτελέσματα από οποιαδήποτε προηγούμενη κρίση. Και αυτό για διαφορετικούς λόγους. Όχι μόνο λόγω της έκτασης της κρίσης που καλύπτει πάρα πολλού φορεί, αλλά και διότι καλύπτει πάρα πολλούς οικονομικούς φορείς και συγκεκριμένα τις αεροπορικές εταιρείες σε μια φάση που ακόμα προσπαθούν να ξεπεράσουν την προηγούμενη κρίση και να αποκαταστήσουν τη θέση τους. Δεν έχουμε βγει λοιπόν ακόμα από την προηγούμενη κρίση και έτσι χτυπάει η νέα κρίση. Όταν βρισκόμασταν στην προηγούμενη κρίση είχαμε μια διαφορετική διάρθρωση της αγοράς όπου η λεγόμενη supply chain, η αλυσίδα προμηθείας ήταν υπό τον έλεγχο μία, της κάθε μίας εταιρείας. Μία από τις απαντήσεις στην προηγούμενη κρίση είναι να υπάρχουν οι λεγόμενοι τρίτη και τέταρτη φορείς οι οποίοι είναι υπεργολάβοι υπηρεσιών για εξοπλισμό και για υπηρεσίες της εταιρείας αυτές. Λοιπόν, η αλυσίδα τροφοδοσίες που συμβάλλει στην παραγωγή του τελικού προϊόντος που είναι οι αεροπορικές μεταφορές έχει επεκταθεί για πολύ περισσότερους εμπλεκόμενους φορείς και επομένως έχει, είχε κινηθεί προς πιο ειδικευμένους τομείς. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά αυξήθηκε και η έκθεση σε κινδύνους των εταιριών και γι' αυτό η κρίση αυτή είναι πιο έντονη γιατί <clears throat> καλύπτει τις αεροπορικές εταιρίες, χτυπάει τις αεροπορικές εταιρείε σε μια φάση ανάκαμψης που δεν έχουν ακόμα επιτύχει μια πλήρη αναδιάθρωση για να αντιμετωπίσουν μια νέα κρίση και επειδή είναι πολύ μεγαλύτερο ο αριθμό των εταιριών οι οποίες φύγονται. Είναι μια κρίση λοιπόν με διαφορετικές διαστάσεις από, την κρίση που είχαμε, από τις κρίσεις που είχαμε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα. Ε, ε, Όσον αφορά τη δεύτερη και τρίτη ερώτηση για τη Μέση Ανατολή και τι συμβαίνει. Πήγαμε και οι δύο στο Αμπού Ντάμπι πριν από κάποιους μήνες. Και εκεί διαπιστώσαμε ότι είναι πολύ επιθετική πολιτική προμήθειά τους. Αν δείτε τα προγράμματα των εταιριών τους, όπως είναι η Etihad, παραγγέλουν 50-60 μεγάλα ε, αεροσκάφη, ήδη έχουν πληρωθεί, ευρείας ατράκτου και αυτό τη σωστή στιγμή, άμα γίνει, σκοτώνει τον ανταγωνισμό, κυρίω τον ανταγωνισμό που δεν έχει ρευστό. Αν δείτε ποια είναι η πολιτική των δύο μεγάλων αεροπορικών εταιριών μέσα Μέση Ανατολή, είναι διαφορετική. Η Etihad είναι λιγότερο επιθετική από την Emirates. Αλλά έχει τεράστια υποθέματα ρευστού. Και έχει στεγνώσει το ρευστό τη Emirates. Και στο μέλλον ίσω αλλάξουν. Αλλά βλέπετε αυτή την αλλαγή όσον αφορά και τους κόμβους προς τη Μέση Ανατολή, Αμπού Ντάμπι και Ντουμπάι και το Κατάρ σε κάποιο βαθμό, θα δείτε ότι εκεί οι συνέπειες είναι πολύ μεγάλες. Συγκέντρωση. Είπατε ότι υπάρχουν τρεις μεγάλοι, μεγάλα πλέγματα στην Ευρώπη. Είπατε πόσες συμμαχίες μπορούν να, συμμαχ... να επιβιώσουν. Αλλά δείτε, στην Αμερική έχουμε τρεις μεγάλες εταιρείες. Τι βλέπετε. Βλέπουμε ομαδοποιημένα στοιχεία για αυτές τις συμμαχίε, αλλά εκεί κρύβονται πολλά πράγματα. Αν θες να κυριαρχήσεις, μπορείς να κυριαρχήσει σε κάποια δρομολόγια κάτω από κάποιες συνθήκες στα πλαίσια κάποιες συχνότητες δρομολογίων. Ίσως μπούμε σε λεπτομέρειες σε αυτό το θέμα αργότερα, αλλά θα απαντήσουμε με τη σειρά στις ερωτήσεις. Για τις χρονοθυρίδες, ο πρόεδρος ζητάει συντομία είναι μεγάλος, γιατί είναι μεγάλος ο κατάλογος αυτών που θέλουν να λάβουν το λόγο. Για την διαταραχή που προήλθε σε σχέση με τα σλότς. Εδώ φαίνεται πραγματικά και η τροποποίηση του ρόλου του αεροδρομίου που περνά από μια παθητική υποδομή στο να γίνεται μια ενεργητική υποδομή που έχει ένα προϊόν να πουλήσει. Και το προϊόν αυτό είναι το σλότ, η χρονοθυρίδα. Αυτή ήταν μια ριζοσπαστική αλλαγή στην στον αεροπορικό κλάδο και στα αεροδρόμια. Από την άποψη αυτή, η αναγνώριση της ύπαρξης ενός εμπορικού προϊόντος από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και η κάλυψή του από την ρύθμιση είναι κάτι το οποίο θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα θετικό. Τα άλλα δύο ερωτήματα τώρα. Λοιπόν, κοιτάξτε. Πώς μπορεί κανείς να μετρήσει τη συγκέντρωση. Νομίζω ότι είναι θέμα στρατηγικής συμπεριφοράς. Το βλέπει κανείς στις θαλάσσιες μεταφορές. Βλέπεις τα μερίδια της αγοράς και μπορείς να σχηματίσεις για κάποιες διαδρομές τι γίνεται. Βλέπεις συχνότητα δρομολογίων, και κυρίως εξετάζεις και την τιμολόγηση και βλέπεις πώς καθορίζονται οι τιμές. Ρωτήσατε τι γίνεται με την αγορά των εταιριών χαμηλού κόστους. Πάνε καλύτερα τα πράγματα από ό,τι αλλού ή όχι. Η απάντηση είναι όχι. Αν θέλετε προσωπική άποψη, δεν το λέει αυτό το έγγραφο, όσο με αφορά, αν δείτε το μοντέλο της Ryanair, εκεί βλέπετε ότι υπάρχουν προβλήματα. Τα νέα μοντέλα που, αγοράζονται και δεν πληρώνονται λοιπά δημιουργούν προβλήματα. Η κυρία Φώστερ, ναι, αν είναι η χειρότερη κρίση ή όχι. Δεν ξέρουμε αν δεν τελειώσει η κρίση. Ρωτήσατε και το θέμα των εμπορευμάτων, τι γίνεται με τη μεταφορά εμπορευμάτων. Αν δείτε τι γίνεται σε 30 χρόνια στην αγορά, βλέπετε ένα κενό το 2001 και μετά το 2001 ο συντελεστής ανάπτυξης ήταν περίπου ο ίδιος όπως ήταν πριν το 2001. Δεν συμφωνούμε κατά πόσο ο ρυθμός ανάπτυξης θα είναι ο ίδιος μετά την μεγάλη πτώση 2008-2009. Με ρωτήσατε τι θα κάνουμε δεν είναι η πρωτογενή ζήτηση, η δευτερογενή ζήτηση για μεταφορέ είναι αυτή που υπάρχει. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντιρόν πρώτη. Είναι η επόμενη τώρα στάδα ερωτήσεων. Τη ερωτήσει ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή η μελέτη ήρθε ακριβώ στη σωστή ώρα, πριν από τη Σύνοδο Κορυφή τη Κοπενχάγη, πριν από τη συζήτηση επί τη Λευκή Βίβλου που επίκειται. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη και θα τη διαβάσουμε λεπτομερώς. Δύο σύντομες ερωτήσεις έχω αφορούν το θέμα της συγκέντρωσης ουσιαστικά. Κανονικά επιτρέψτε μου να πω, δεν είμαι οικονομολόγος, κάποιος απλοϊκή ερώτηση, αλλά θεωρούσα ότι η απελευθέρωση του τομέα είχε σαν στόχο πάνω απ' όλα να επιτρέψει να ξεφύγουμε από τα δημόσια μονοπόλια και να έχουμε μεγαλύτερο ανταγωνισμό και να έχουμε πολυπληθείς φορείς στον ιδιωτικό τομέα και καταλήγουμε σε ιδιωτικό μονοπόλιο ή σε μεγάλα ιδιωτικά μονοπόλια ακόμα αν είναι κατά περιοχή του κόσμου, ε, κατά διαδρομές, υπάρχουν ε, κάποιες κατανομές αγοράς και μας δώσατε κάποιες συστάσεις και μας εξηγήσατε τι γίνεται με την παρακολούθηση και τον έλεγχο. Δεν μας λέτε όμως τι θέλουμε σαν μοντέλο. Θέλουμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της αγοράς που κινείται προς συγκέντρωση, ακριβώς το αντίθετο που θέλαμε απευθύνοντας την αγορά. Θέλαμε τις μικρές εταιρείες να τις πολλαπλασιάσουμε, να υπάρχει ανταγωνισμός, να βελτιώσουμε την ποιότητα, να έχουμε καλύτερες τιμές για τους επιβάτες για εκείνους που μεταφέρονται. Είναι σύνηθε να διαπιστώνεται απλώς ότι υπάρχει συγκέντρωση. Δεν θα ήταν πιο χρήσιμο να διαρωτηθούμε τι μοντέλο θέλουμε για τη μικρή απόσταση, τη μέση απόσταση, τη μεγάλη απόσταση όσον αφορά τις μεταφορές και να προσπαθήσουμε να προσανατολίσουμε την αγορά παρά να τρέχουμε πίσω από την αγορά. Ενώ τα αποτελέσματα της απελευθερώσεως είναι τα αντίθετα από αυτά που είχαμε ανακοινώσει. Αυτό είναι ένα γενικό ερώτημα που σας υποβάλλω. Αντιπρόεδρος Ρίκε. Κοιτάξτε, ήθελα να κάνω την μία διαρώτηση με τον Ματίας Προηγουμένος. Δεν απαντήσατε σε μία ερώτηση που αφορά τα σλότ. Αν υπάρχουν ε, μέτρα τα οποία εξέπνεαν ε, στις 30 Οκτωβρίου και ουσιαστικά θα υπάρξει μία νέα νομοθεσία ε, λόγω, ώστε, ώστε να αναβληθούν... Ε, να μην υπάρξουν όλες αυτές οι αρνητικές συνέπειες από την νομοθεσία τη σχετική με τα σλότ, γιατί την ερώτηση την έθεσε και ο συνάδελφος προηγουμένως. Μου φαίνεται ότι το μέτρο αυτό σταματούσε να ισχύει στις 31 Οκτωβρίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη γιατί το έχουν αναφέρει πολλοί από τους συναδέλφους ήδη προηγουμένως. Αυτή τη στιγμή, μέσω αυτής της κρίσης, βλέπουμε ότι πάρα πολλές μορφές μεταφορών έχουν πληγεί, όχι μόνο οι μεταφορές. Πιστεύω ότι φτάσαμε στο χαμηλότερο σημείο και τα πράγματα τώρα πάνε κάπως καλύτερα. Ελπίζουμε ότι αυτό ισχύει και για την εμπορευματική μεταφορά και για τις επιβατικές μεταφορές. Αυτό το οποίο θα θέλαμε να ξέρουμε είναι ποια είναι η κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Λέτε ότι εκεί πέρα υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα και μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών εκεί. Εμεί θα θέλαμε να έχουμε ένα λειτουργικό σύστημα ανταγωνισμού μέσα στις, ε, στην Ευρώπη και με εταιρείε οι οποίες θα είναι και χαμηλού κόστους ακόμα, αλλά δεν θέλουμε οι ευρωπαϊκές εταιρείες να χάσουν σε σχέση με τους ανταγωνιστές σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν είναι οι επιδοτήσεις η λύση, αλλά κατά τα άλλα εσείς τι προτείνετε για να γίνει στην Ευρώπη για να αντιμετωπίσουμε τις εταιρείε όπως είναι η Emirates, η Etihad, οι οποίες μπορεί να αγοράζουν μερίδια αγοράς και να κάνουν δύσκολη τη ζωή των ευρωπαϊκών εταιρεών. Έχετε κάποιες ιδέες ή έχετε κάποιες, ε, ε κάποια αιτήματα από εμάς Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ένα σχόλιο και μία ερώτηση. Νομίζω ότι αυτή η έκθεση είναι κάπως αεροπορικό εταιρείο κεντρική σε ό,τι αφορά τις απώλειες θέσεων εργασίας, γιατί υπάρχει και ο ευρύτερο τομέα της αεροπορίας όπου χαθήκανε θέσεις εργασίας. Η ερώτηση ήταν ποιος είναι ο ο αντίκτυπος της κρίσης σε όλο τον τομέα των αεροπορικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μονάχα στις αεροπορικές εταιρείες όπου έχετε εστιάσει την προσοχή σας. Αυτό είναι απλώς ένα σχόλιο. Το ερώτημά μου, ίσως είναι αμφιλεγόμενο αυτό το οποίο λέω, αλλά με ενδιαφέρει η απάντησή σας. Από ό,τι έχω ακούσει, και πάλι δεν έχω διαβάσει την έκθεση, την είδα μαζί με τους άλλους βουλευτές εδείς. <clears throat> Υπάρχει κάποιος κίνδυνος η Lufthansa και η Star Alliance να αποκτήσουν μια δεσπόζουσα θέση στην Ευρώπη και να χρησιμοποιήσουν αυτή την κρίση για να αποκτήσουν μια δεσπόζουσα θέση ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Okay. Um, ehm, de vraag van, van mevrouw Ωραία, θα απαντήσω στην κυρία Durand πρώτα. Κατανοώ τα επιχείρηματά σας ότι η φιλελευθερωποίηση έγινε με τον τρόπο που περιμέναμε. Και από αυτή την άποψη μπορώ να συμφωνήσω μαζί σας. Αυτό όμως το οποίο συμβαίνει τώρα είναι ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο μόνο στον τομέα της αεροπορίας, αλλά και σε άλλους τομείς. Είδαμε λοιπόν ότι εκπληρώθηκαν οι προσδοκίες μας στον τομέα αυτό. Ίσως μπορούμε στο μέλλον να διορθώσουμε την πορεία που έχουν λάβει οι τομείς αυτής. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο περιέχεται στα βασικά εγχειρίδια βιομηχανικής οικονομίας και βιομηχανικής πολιτικής. Το ερώτημα είναι πότε θα βρούμε την κατάλληλη στιγμή για να επέμβουμε, πώς θα πρέπει να μελετήσουμε την προβληματική για να βρούμε τα καλύτερα μέτρα τα οποία χρειάζεται. Και σε σχέση με κάποια άλλα ερωτήματα, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι έχουμε ενώπιόν μας μια κρίση η οποία μας κατέλαβε όλους εξαπίνης. Το ερώτημα πώς θα μπορέσουμε λοιπόν να αναλύσουμε αυτή την κατάσταση και να δούμε αν υπήρχαν κάποιοι δείκτες οι οποίοι ήδη μας έδιναν πληροφορίες για να προβλέψουμε την κρίση. Αυτή τη στιγμή όμως δεν έχουμε κανένα τέτοιο δείκτη. Νομίζω θα ήταν πρόωρο να προσπαθήσουμε να δούμε αν υπήρχαν κάποιες τέτοιες ενδείξεις στο παρελθόν. Έχουμε λοιπόν κάποιες ε, ιδέες, αλλά δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα γίνει στο, στο μέλλον. Για τα slots, νομίζω ότι το βασικό ε, ερώτημα είναι το use it or lose it. Χρησιμοποιήστε τα ή χάστε τα. Αυτός ο κανόνας σε εποχές κρίσης δίνει μια μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Γιατί πολλές φορές οι χρονοθυρίδες χρησιμοποιούνται για να μπλοκάρουν την αγορά, όχι να την αναπτύξουν. Υπάρχει μια μακρά εμπειρία στην, στον αεροπορικό κλάδο για τη χρήση μιας τέτοιας στρατηγικής. Όταν έχουμε μια κρίση, οι εταιρείε δεν έχουν οικονομικούς πόρους για να εφαρμόσουν μια στρατηγική μπλοκαρίσματος των σλότ. Επομένως, αυξάνει η αποτελεσματικότητα της χρήσεως ε, αυτού του εργαλείου των σλότ. Πρέπει να διατηρήσουμε τα σλότ γιατί είναι πράγματι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο ελέγχου της βιομηχανίας. Έχει περάσει η κρίση τώρα. Εγώ προσωπικά πιστεύω όχι, ότι δεν έχει ξεπεραστεί η κρίση. Αυτή τη στιγμή εμείς εξετάζουμε τους δείκτες σε καθημερινό επίπεδο, σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές και τις εναέριες μεταφορές. Μερικές φορές φαίνεται ότι ένας δείκτης έχει φτάσει στο χαμηλότερο σημείο και αρχίζει να ανέρχεται, αλλά δεν συμβαίνει αυτό πάντα. Σε ό,τι αφορά τους σταθερούς δείκτες δεν νομίζω ότι υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή για κάποιο χρονικό διάστημα είχαμε την εντύπωση ότι τα πράγματα επανερχόντουσαν, ότι υπήρχε ανάκαμψη, αλλά αυτό είναι σαν το να υπολογίζει κανείς σε Χριστουγεννιά τους μπουναμάδες προτού τους πάρει. Τώρα, το ερώτημα του τι θα γίνει με τα κεφάλαια των εταιριών και τα αποθεματικά που έχουν σε κεφάλαιο. Εγώ ήμουν σε επαφή με ένα εκπρόσωπο της Etihad, και η επιχείρηση αυτή δίνει μεγάλη σημασία στην δομή των κεφαλαίων σε αυτή την επιχείρηση. Αυτό δεν είναι καινούριο. Εδώ και πέντε, εδώ και 10 χρόνια πολλές από τις επιχειρήσεις στον αεροπορικό τομέα στην Ευρώπη ήδη είχαν αρχίσει να βλέπουν τι κάνουν οι ομολογοί τους, οι Singapore Airlines, οι Μαλέσια, μαζεσιανές αεροπορικές γραμμές. Επομένως, κοιτάνε με ποιο τρόπο λειτουργεί αυτή η αγορά. <clears throat> Το ερώτημά σας λοιπόν είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλλά έχουμε ένα αποτέλεσμα ασυγχρόνου χαρακτήρα. Αυτό το οποίο συμβαίνει ότι οι εταιρείε οδηγούν σε μια απώλεια θέσεων απασχολήσεως, όπως ελέγχθη, αλλά αυτές οι απώλειες θέσεις απασχόλησης οδηγούν σε νέες οικονομικές δραστηριότητες. Βλέπουμε λοιπόν τι γίνεται στην αεροπορική βιομηχανία με την δημιουργία των forwarders στις ε, επίγες, στις χερσαίες μεταφορές. Λοιπόν, αργά ή γρήγορα, το κύμα της κρίσης και το κύμα των ε, απολύσεων ξεπερνιέται και επομένως θα έχουμε την ε, απώλεια θέσεων απασχόλησης στους άλλους φορείς οι οποίοι συνδέονται με τις αεροπορικές εταιρείες. Αυτή τη στιγμή όμως δεν έχουμε συγκεντρωμένες πληροφορίες για να μπορούμε να ξέρουμε ποιο είναι το επίπεδο ανεργίας στις εταιρείες αυτές και επομένως το πώς θα διαχυθεί η ανεργία μέσα στην λυσίδα προμήθειας των εταιριών. Το τελευταίο ερώτημα ήταν η δεσπόζουσα θέση της Θαραλάνης και της λουκάς. Λοιπόν, όσον αφορά αυτό το θέμα, θα έχουμε αυτές τις τρεις μεγάλες συστάδες και θεωρητικά θα πρέπει να εξισορροπούνται. Ε, στο κάτω-κάτω είναι προς όφελός τους να γίνει αυτό. Και υπάρχει ένα φαινόμενο. Ας πάρουμε τη Star Alliance. Ας μην θεωρηθεί σαν ομοιογενής αυτή η Star Alliance. Υπάρχει εσωτερικός ανταγωνισμός εντός της Star Alliance. Αν θες να πας από τη Βρυξέλλες στο Σικάγο, Μπορείς να πας μέσω Φραγκφούρτης, από Βρυξέλλες Σικάγο, ή να πάει στη United και να πας μέσω Washington. Αυτός είναι εσωτερικός ανταγωνισμός μεταξύ δύο εταιριών εντός της συμμαχίας, Lufthansa και United, εντός της Star Alliance. Θα εξακολουθεί να υπάρχει ο ανταγωνισμός από τη στιγμή όπου δεν υπάρχει απόλυτη κυριαρχία εντός μίας από τις τρεις μεγάλες αυτές εναπομένουσες συμμαχίες. Εγώ ανησυχώ ότι μπλοκαρίστηκε λόγω δεσπόσα θέση το θέμα αυτό με την ε, BAA και ενώ η Star Alliance αρπάζει χρονοθυρίδες από κάθε αεροδρόμιο και μαζεύει και όλα τα αεροδρόμια. Εκεί υπάρχει ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που παρουσιάσατε την έκθεσή σας, ευχαριστώ που απαντήσατε στις ερωτήσεις των μελών και αν τα μέλη έχουν και άλλες ερωτήσεις όταν διαβάσουν το κείμενο, είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν σε επαφή μαζί σας και ελπίζω ότι θα τους δώσετε κάποια απάντηση. Ευχαριστώ. Πριν εξαφανιστούν τα μέλη, κύριε Αλκαντράουι, έχουμε κάποια σημεία στα διάφορα. Έχω, έχω. Η κυρία Φώστερ έχει κάτι στα διάφορα και ο πρόεδρος έχει κάτι στα διάφορα. κυρία Φώστερ, μην τους αφήνετε να φύγουν τόσο νωρίς. Λοιπόν, το έχω θέσει ξανά το θέμα αυτό, διότι αφορά τα, τους εκλογείς και εστιάζεται περισσότερο στους Ισπανούς φίλους μας και αφορά τους οδηγούς φορτηγών. Και τι συμβαίνει. Δεν μπορώ να ακούσω, μιλάνε, συζητάνε, τάξη, τάξη, ησυχία. Δεν θέλω να διαβάσω όλη την επιστολή. Λοιπόν, δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τους Βρετανούς οδηγούς φορτηγών αλλά και άλλους. Όταν είναι στην Ισπανία λοιπόν οι οδηγοί των φορτηγών σταματήστηκαν και τους επευλήθησαν πρόστιμα χιλιάδων ευρώ κάτι με τον ταχυγράφο, κάποιο πρόβλημα ταχυγράφο. Δεν μπόρεσαν να μετακινηθούν έως ότου πληρώσει το πρόστιμο. Και όταν ελέγχθηκαν αργότερα όλοι οι ταχυγράφοι είδαν ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα όταν έγινε ο έλεγχος από τους αρμόδιους φορείς. Συχνά συμβαίνει αυτό φαίνεται. Δεν υπάρχει διαδικασία εφέσης, ήρθαν σε επαφή με τη Βρετανική Πρεσβεία να τους πούν τι, κάνουν, τι μπορούμε να κάνουμε, ρωτήσαμε μας ζητάνε χιλιάδες ευρώ. Και φαίνεται ότι είναι μεγάλο πρόβλημα και το θέτω εδώ στην Επιτροπή διότι θεωρώ ότι εσείς ε, σαν πρόεδρος μπορείτε να το εξετάσετε μπορούμε να δούμε κατά πόσο είναι πιο ευρέω διαδεδομένο το φαινόμενο. Και με του Ισπανού συναδέλφου μπορούμε να κάνουμε κάτι, να ερευνήσουν οι Ισπανοί συνάδελφοι, γιατί θα πρέπει να υπάρχουν ισότιμε συνθήκε όσον αφορά τα φορτηγά μα που ταξιδεύουν σε όλη την Ευρώπη. Και νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αν μας δώσετε λεπτομέρειες, αν δώσετε λεπτομέρειες στην γραμματεία, εγώ θα ετοιμάσω μία επιστολή και θα στείλω μία επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντα κάποια εξήγηση από τον αρμόδιο επίτροπο. Και ίσως ε, να αποσταλεί και αντίγραφο στην μόνιμη ισπανική αντιπροσωπεία που έχουν και την Προεδρία από 1η Ιανουαρίου. Λοιπόν, δώστε λεπτομέρειες στη γραμματεία για να ετοιμάσουμε την δέουσα επιστολή. Το δεύτερο που έχω αναθέσει εδώ, να υπενθυμίσω στα μέλη ότι θα διεξαχθεί μια συζήτηση όταν αφορά την πειρατεία στις θάλασσες με τον υπονάβαρχο Χότσον στη συνάντηση Επιτροπής ΕΝΤΕΣ της 16 Νοεμβρίου στις 3. Τα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν στην ανταλλαγή απόψεων. Ένα μέλος της Επιτροπής μας πήγε στα αρχηγείο των μεικτών επιχειρήσεων όταν πήγε η Επιτροπή ΣΕΝΤΕ και μα προσκάλεσε η Επιτροπή αυτή σε... επειδή καλέσαμε τον επικεφαλής αξιωματικό και τον υπαρχηγό, νομίζω ότι είναι Γάλλος Ναύαρχος, να έρθουν και να μας μιλήσουν στην Επιτροπή, προσεκλήθημεν και εμείς, στις 3-16 Νοεμβρίου. Πειρατεία στις θάλασσες. Αν οι συντονιστές σας ενημερώσουν τα μέλη των ομάδων. Υπάρχει άλλο θέμα στα διάφορα. Εάν δεν υπάρχει άλλο θέμα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διερμηνείς για τη δουλειά τους, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εκείνους που απουσιάζουν τώρα και που είχαμε σε αυτή τη συνεδρίαση, όχι μόνο διερμηνείς, αλλά και διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας για έναν βουλευτή. Ευχαριστώ όλους τους διερμηνείς, είτε χρησιμοποιούν φωνή, είτε νοηματική γλώσσα για τη δουλειά τους και κυρίσω το πέρας της συνεδρία σα. Καλή σας νύχτα. other than has been as a local member.